Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην συνεδρίασή μας, τη συνεδρίαση Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Νομίζω ότι είναι <clears throat> η τρίτη από το τέλος συνεδρίας που θα κάνουμε πριν ολοκληρωθεί η εντολή αυτή. Λοιπόν, ας εγκρίνουμε καταρχάς την μερίσια διάταξη, σημείο 1. Σας προτείνω να κάνουμε εδώ πέρα μία αλλαγή στη μερίσια διάταξη λόγω της απόφασης της διάσκεψης των Πρόεδρων την προηγούμενη εβδομάδα, όπου γίνεται ένα ξεκάθαρο αίτημα να μην ψηφίσουμε καμία έκθεση, ακόμα και επιστολή που να έχει σχέση με το Brexit, σας προτείνω να αναβάλουμε τη συζήτηση που προβλεπόταν στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης, την ψηφοφορία μάλλον που προβλεπόταν στο σημείο 11, σύναψη της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση γνωμοδότηση Γκουίστουλ Τερόφολ. Υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς την προτινόμενη αυτή αλλαγή στη μερίσια διάταξη. Όχι, επομένως εγκρίνεται αυτή η τροποποίηση. Υπάρχουν ε, άλλε προτάσει τροποποίηση τη μερίσια διάταξη. Όχι, επομένω μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Περνάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων τη 23, 23 και 24 η Ιανουαρίου 2019. Το σχέδιο πρακτικών σας έχει διανεμηθεί και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά εγκρίνονται μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Οι αποφάσεις των συντονιστών που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου περιλαμβάνονται στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης. Επομένω, ισχύει και εδώ πέρα ο ίδιο κανόνα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρίαση, θεωρείται ότι εγκρίνονται και αυτέ οι αποφάσει. Σημείο 4 τώρα. Ανακοινώσει του Προέδρου. Ο συνήθω, πρέπει να σα πω ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Επομένω, καλημέρα σε όλου, από όπου και να μα ακούτε, από το Ταλίν, τη Θεσσαλονίκη, από όλε τι γωνιέ τη Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την διερμηνία, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην μιλάνε πολύ γρήγορα, να μιλάνε αργά, να είναι σαφείς, προκειμένου να μπορούν να καταλάβουν και οι διερμηνείς. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Μαριόλα Αλβάρας Λόπες, η οποία κάθεται εκεί, όπως βλέπετε, η οποία εργάστηκε για πολλούς μήνες στη γραμματεία της Επιτροπής μας, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρουμε ότι θα φύγετε από τη γραμματεία. Σας ευχόμαστε καλή τύχη για το μέλλον. Έτσι περνάμε στο σημείο 5 της μερίσιας διάταξης όπου προβλέπεται συζήτηση για την ε, γνωμοδότηση τη Επιτροπή μα όσον αφορά τη σύνοψη της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Λόγω της απόφασης που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίστηκε ότι οι διάφορες κοινοβουλευτικέ επιτροπές που εμπλέκονται στην ε, όλη διαδικασία που έχει να κάνει με το Brexit θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν με τη μορφή επιστολής προς την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή που είναι η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων, η ΑΦΚΟ. Εξαιτίας της επίγουσας διαδικασίας που ακολουθείται, Θεωρώ ότι είναι εντελώ λογικό και εμεί να κινηθούμε έτσι, να γνωμοδοτήσουμε δηλαδή μέσω επιστολή. Λόγω όμω τη απόφαση που ελήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων την προηγούμενη εβδομάδα, όπου αποφασίστηκε εκεί να μην ψηφίσουν ακόμα οι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ για τι επιστολέ αυτέ, προτού αποσαφινιστεί λίγο περισσότερο η όλη κατάσταση και η διαδικασία στην Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Μπορούμε και εμεί να αναβάλουμε λοιπόν, όπω αποφασίσαμε την ψηφοφορία αυτή, και μπορούμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο την εν λόγω επιστολή. Βλέπετε ήδη ότι οι συντονιστέ έχουν συμφωνήσει επ' ενός σχεδίου κειμένου για αυτή την επιστολή, εξαιτία όμω τη ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση σε σχέση με το Brexit ενημερώθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ακόμα έτοιμη ή δεν διατίθεται ή δεν επιθυμεί ακόμα να πάρει το λόγο για το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο τη σημερινή μα συνεδρίασης. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρκετά αυτόνομο και ισχυρό, προκειμένου να μπορεί να σχολιάσει και μόνο το ζήτημα αυτό, χωρί την συμβολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Του τον λεχθέντο να δώσω το λόγο στην εισηγητριά μα. Γκουίστο Λορόβολτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σα ζητώ συγγνώμη που δεν παρευρέθην εδώ από την αρχή της συνεδρίασης στην αίθουσα, οπότε ενδεχομένω να επαναλάβω εν μέρη τα όσα ήδη είπατε. Πράγματι, αναφέρθηκε ότι οι επιτροπές εκείνες οι οποίες είναι συναρμόδιε ε, και μπλέκονται σε αυτές τις πραγματεύσεις του Brexit καλό θα ήταν να αποτυπώσουν την άποψή του σε μια γνωμοδότηση. Και καθώ εργαζόμαστε πάντοτε υπό την πίεση χρόνου σε αυτό το κοινοβούλιο και σε αυτή την περίπτωση ε, αποφασίστηκε ακριβώς λόγω της πίεσης χρόνου να συνταχθεί μια επιστολή και αυτή η επιστολή αφορά ε, κυρίως ε, τις επιτροπές ΑΦΕΤΕ και ΕΝΒΗ. Τώρα το κατά πόσο έχουν αποφασίσει και άλλες επιτροπές να συμμετάσχουν δεν το γνωρίζω. Η κατάσταση δηλαδή που σας περιγράφω ίσχυε την προηγούμενη εβδομάδα ε, χθες το βράδυ στις 7.30 έλαβα ένα τηλεφώνημα όπου μου ζητήθηκε να μην λάβει χώρα αυτή η ψηφοφορία. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη μας ε, το γεγονός ότι έχει συνταχθεί μια επιστολή, αλλά ακόμα να μην ψηφίσουμε μέχρι να έχει διαμορφώσει η Επιτροπή ή το Συμβούλιο, δεν ξέρω ποιο, μία άποψη. Τουλάχιστον αυτό μου ζήτησαν τηλεφωνικώ. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, αλλά ας μην προβούμε σε ψηφοφορία. Ε, αυτό που απήντησα χθε είναι και αυτό που θα πω ε, εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω τι σχέση έχει η ΑΦΚΟ και ποια αρμοδιότητα ε, έχει η ΑΦΚΟ για αυτή την περίπτωση ε, όταν έχουμε να κάνουμε μια χώρα η οποία στον κείμενο δεν θα περιλαμβάνεται πλέον ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν νομίζω πως έχει φτάσει η χρονική στιγμή όχι μόνο να εστιάσουμε στο withdrawal agreement, δηλαδή στη συμφωνία αποχώρησης, αλλά και στο τι θα ακολουθήσει μετά από την λόγο ε, συμφωνία και νομίζω πως η δική μας Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ε, είναι πολύ πιο αρμόδια από οποιαδήποτε άλλη περισσότερο διαχειριστικού αν θέλετε χαρακτήρα Επιτροπή. Οπότε, εντάξει, αυτή ήταν δική μου άποψη και από εδώ και μετά δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ πρότεινα ενδεχομένως να συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά ε, την, ε, το σχετικό ψήφισμα του Συμβουλίου ή από την άλλη πλευρά μπορούμε να ε, αναμείνουμε με την δική μας ψηφοφορία για να δούμε τι θα κάνουμε. Πρόεδρος, ναι, Κοντελίβε, ήδη κατά την έγκριση της ημερής σας διάταξης αποφασίσαμε ότι θα αναβάλουμε την εγώ ψηφοφορία. Πάντως, συμφωνώ μαζί σου ως προς το ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το ζήτημα δεν είναι ιδιαίτερα διαφανής και δημοκρατικός. Ε, και αυτό και, και διαλέγω προσεκτικά εδώ τα λόγια μου. Η διάσεψη των Προέδρων έλαβε την ελόγω απόφαση την περασμένη εβδομάδα την περασμένη Πέμπτη, ε, δηλαδή του να είναι ανεξάρτητες ε, ε, οι γνωμοδοτήσεις και τοποθετήσεις των επιτροπών εντελώς ανεξάρτητε είναι κάτι με το οποίο ε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή πραγματικά εκείνο που κάναμε μέχρι τώρα και ήταν η κανονική πρακτική είναι να ε, προσανατολίζονται οι υπόλοιπε επιτροπές ε, στην τοποθέτηση του leading κομμάτι της αρμόδιας δηλαδή επί τη ουσία επιτροπής για μια χρονοδότηση. Αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο συνάδελφο που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ο κύριος Σούστα. Ναι. Ε, αρχίζει σιγά σιγά να με ανησυχεί η κατάσταση που επικρατεί. Γιατί πράγματι ισχύει ότι η Βρετανική κυβέρνηση έχει αποτύχει πλήρως ε, γιατί δεν έχει ούτε καν ένα σχέδιο κατά νου ως προς το πώς θα ήθελε να διαμορφώσει τον Brexit της. Και από εκεί και μετά Ε, αφού δεν ξέρει τελικά πού θα καταλήξει το ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο, τότε ο κύριο Τούσκ είναι εκείνο ο οποίο καλείται να προβληματιστεί περισσότερο. Πάντω, εκείνο που ισχύει είναι ότι βρισκόμαστε ενώπιον ενό σοβαρού προβλήματο. Ετούσκη δηλαδή, ειναι όλοι λένε ότι θέλουμε να λάβει η χώρα με τακτικό τρόπο, με οργανωμένο τρόπο το Brexit και όλοι λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει σκληρό σύνορο μεταξύ Ιρλανδίας και Βορείου Ιρλανδίας, αλλά τελικά έτσι όπως τα πράγματα διαμορφώνονται θα υπάρξει αυτό το σύνορο. Γιατί όταν ρωτάμε τη Βρετανική κυβέρνηση ως προς το πώς θέλει να διαμορφώσει αυτήν την ε, αυτό το, το, την μη ύπαρξη αν θέλετε σε σκληρό συνόρο, εάν δεν υπάρξει συμφωνία Brexit, ε, βλέπουμε ότι δεν έχει κάποια απάντηση να μα δώσει. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων θα οδηγηθούμε σε σκληρό σύνορο. Και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω περισσότερα επί τις διαδικασίες. Δηλαδή τι κάνουμε αυτή την ε, περίοδο. Το Συμβούλιο δηλαδή και η Επιτροπή ε, προσπαθούν να οργανώσουν τα πράγματα από τη δική τους πλευρά και εμεί το μόνο που κάνουμε από πλευρά του Κοινοβουλίου για να μην περιέλθουμε σε δυσκολίες αποστέλουμε απλώ και μόνο μία επιστολή. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, τα πράγματα και οι διαπραγματεύσει θα λάβουν χώρα και κλεισμένων των θύρων σίγουρα θα πρέπει να προβληματιστούμε σοβαρά ως προς το τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ε, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορο στο πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα στο πλαίσιο του Brexit στο μέλλον. Και εμά μα ενδιαφέρει πολύ. Άρα λοιπόν θα ήθελα να ακούσω. Λαμβάνουν χώρα έστω και παρασκηνιακά διαβουλεύσει. Και αν όχι, ε, κατά την επόμενη όλο μέλη θα πρέπει να το αξιώσουμε αυτό κατηγορηματικά. Δηλαδή να μην υπάρχουν επιμέρους θεσμικά όργανα τα οποία έρχονται σε διάλογο ε, με την ε, Βρετανική πλευρά χωρίς να υπάρξει μια συντονισμένη εδώ τοποθέτηση από την πλευρά ε, και τη δική μας. Και έχουμε και τους, απόλυτους, τους ραζίτικους εκπροσώπους από τη δική μας πλευρά. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, ο κύριος Σόλς. Ναι, νομίζω πως όλους μας ανησυχεί και μας δημιουργεί πραγματικές ανησυχίες αυτή η κατάσταση. Πάντως, δεν είναι το ζητούμενο εδώ το κατά πόσο είναι αρμόδια όχι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Το εκείνο που μας προβληματίσει είναι το ότι ε, το γεγονός ότι ε, ήδη όλα τα μέλη εκείνης της Επιτροπής έχουν τώρα γίνει ε, μέλη και της σχετικής διαχειριστικής επιτροπής με αποτέλεσμα βέβαια να, αλλάβει, ακόμα ε, περισσότερο αρμοδιότητα, αν θέλετε, περισσότερη σημασία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μας απασχολήσει ε, το, η μελλοντική σχέση που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 πλέον με το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί και σε σχέση με αυτό το ζήτημα υπάρχει ευθύνη που μας βαρύνει σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση αυτής της μελλοντική σχέσης. Άρα λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να προτείνω είναι να εκφράσουμε με σαφήνεια τη δική μας θέση απέναντι στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, δηλαδή θα πρέπει να ε, διαμορφώσουμε με σαφήνεια την άποψή μας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να αναμένουμε ε, έως τις 29 Μαρτίου. Δηλαδή, ε, νομίζω πως αναμένουμε πλέον ότι τα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις και τη μελλοντική γενικότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ένα αμφιβόλο και ενδεχομένως και μέσα σε μια τέτοια επιστολή θα μπορούσαν να αρχίσουν να αποσαφηνίζονται. Εντάξει, ίσως αυτό το ζήτημα να αφορά περισσότερο τους συντονιστές, αλλά αφού το συζητάμε εδώ τώρα, το αναφέρω ότι δηλαδή ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει αύριο αυτή η συνεννόηση με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελα να πάρουν το λόγο. Δεν βλέπω να υπάρχει κανεί. Και από χρονική άποψη, βέβαια, βρισκόμαστε ενώπιον μια τεράστια ε, πρόκληση. Δηλαδή, μία ακόμα ολομέλεια μα απομένει πριν από τον Brexit. Την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου, αν ε, δεν απατώμε. Και έτσι οι δυνατότητε μιας επίσημος υπογραφή τη συμφωνία του Brexit ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά περιορισμένε. Και θα πρέπει όμως να διασφαλιστεί η δημοκρατική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία όσο κι αν ε, ε, βασική αν θέλετε <clears throat> πολύ στοιχειώδη είναι αυτή. Και βέβαια, εδώ θα πρέπει να κληθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί όχι μόνο σε σχέση με τη Συμφωνία για τον Brexit, αλλά και σε ό,τι αφορά μια μελλοντική σχέση. Εάν πράγματι τα καταφέρουμε να κυρωθεί μια τέτοια συμφωνία αποχώρηση, θα ακολουθήσει άμεσα μια εντολή διαπραγματευτική, πρέπει να ακολουθήσει άμεσα μια διαπραγματευτική εντολή για την διαμόρφωση της μελλοντική σχέση. Γιατί θα έχουμε μια μεταβατική περίοδο 21 μηνών για την διαμόρφωση αυτής της ε, μελλοντικής σχέσης, πράγμα το οποίο είναι αρκετά δύσκολο και αποτελεί και εκείνο μια πρόκληση. Είδατε πόσα χρόνια χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε με τον Καναδά και τώρα λέμε ότι σε 21 μήνες θα έχουμε καταφέρει όχι μόνο να καταλήξουμε σε συμφωνία αλλά και να την κυρώσουμε. Αυτό σημαίνει ε, με τη σειρά του ότι θα πρέπει ταχύτατα να δοθεί η διαπραγματευτική εντολή ε, και θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε το δικό μας ρόλο ως Επιτροπή. Και αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πράγματι εμείς ως ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχουμε μεγάλη αρμοδιότητα εδώ. Και στη διάσκεψη των Προέδρων τέθηκε εδώ αυτό το ερώτημα, ότι δηλαδή ποια είναι επί της ουσίας τελικά αρμόδια επιτροπή σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit και ο πρόεδρος είπε έτσι αυθόρμητα αν θέλετε ότι η δική μας επιτροπή είναι η αρμόδια. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι και αποδεκτή αυτή η, ε, ο τρόπος εργασίας των διαφορετικών επιτροπών οι οποίες ε, εργάζονται απομονωμένα η μία από την άλλη. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Γκοντελίβε, έχεις και πάλι το λόγο. Ναι, νομίζω πως υπόθηκαν τα πάντα. Δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι ακόμα. Και ο συνάδελφός μας εδώ που συμμετέχει και στις εργασίες της θα μπορούσε να κάνει ένα ε, ερώτημα εκεί, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ούτε από την άλλη πλευρά μπορούμε να επιβάλλουμε στους Βρετανούς το να δράσουμε τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άρα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση είναι ακριβώς να συντάσσουμε και να αποστέλουμε αυτές τις μίνι επιστολές. Καλώς λέω, ο Πρόεδρος, κλείνουμε και με αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των ομάδων. Er-, ναι. Είχαμε δύο ομάδες, η μία ε, που είχε συζητηθεί σε ό,τι αφορά το, την Μερκοσούρ και η άλλη σε ό,τι αφορά τις χώρες των Άνδεων. Τώρα σε ό,τι αφορά την Μερκοσούρ η σχετική συνάντηση έλαβε χώρα στις 29 Ιανουαρίου με την ε, Σάντρα Καλίνα σε ό,τι αφορά το πού βρισκόμαστε σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Ο κύριος ε, Σαλαφράγκα είναι ο μόνιμος συζητητής μας ε, για αυτό το ζήτημα, αλλά δεν παρευρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Eh, Ευχαριστώ. Η ομάδα παρακολούθησης ε, εξέτασε πολύ προσεκτικά τις δυσκολίες που υπάρχουν στις τελικές φάσεις, στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων, αν μπορούμε να την πούμε έτσι. Εγώ έμεινα με την εντύπωση ότι οι προσδοκίες είναι αρκετά αρνητικές. Οι τελευταίες ε, παράμετροι που συζητήθηκαν ε, δείχνουν ότι δεν υπάρχουν οι για να υπάρξει επαρκής πρόοδος το συμπέρασμά μου είναι πως αυτή την περίοδο θα, της θητείας του Κοινοβουλίου θα είναι δύσκολο να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω αν η Επιτροπή που είναι εδώ παρούσα μπορεί να μας δώσει κάποιες ε, πιο πρόσφατες πληροφορίες για το τι έγινε στο Monitoring Group. Ο Χέρμουτ έχει το λόγο και μετά η Ναι, συμπληρωματικά να πω ότι η ε, Μακουλάτο το ανέφερε πολύ εύστοχα, ότι δηλαδή οι διαπραγματεύσει είναι πάρα πολύ περίπλοκες, υπάρχουν ε, μία σειρά από σημεία τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά και τα ε, GI, τις ε, γεωγραφικές ενδείξεις, αλλά και τα ζητήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας και ειδικότερα της κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Ε, και μετά βέβαια τίθεται και το ερώτημα των συγκεκριμένων αποστόσεων στο πλαίσιο της εμπορικής ε, πολιτικής. Ε, πάντως ε, το επιβεβαιώσαμε και στην ομάδα παρακολούθησης και επιβεβαιώθηκε από πολλούς συναδέλφους το ότι παρά τη συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο για την βιώσιμη ανάπτυξη και τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση των ε, σχετικών ε, υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δράση η ίδια, δηλαδή ενέργειες ορισμένων χωρών της Μερκοσούρ έρχονται σε αντίθεση με αυτό το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε πραγματικά και εμείς από την πλευρά της NGL οφείλουμε να πούμε ότι ε, ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας ουσιαστικά θέλει να ε, επιστρέψει σε επίπεδα εκπομπών ε, το οποίο ίσχυε κατά την περίοδο που είχε τερματιστεί η δικτατορία σε εκείνη τη χώρα που θα σήμαινε δηλαδή δεκαπλάσια ουσιαστικά επίπεδα σε συνάντηση και με τα όσα τελικά κάνει δηλαδή σε, σε επίπεδο μόλις η βιομηχανία ειδικότερα στο βορρά της χώρας. Οπότε πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τις χώρες της Μερκοσούρ ή την Βραζιλία ως μοναδικό ως μοναδική χώρα, αλλά έχει να κάνει με, την, ε, με αυτόν τον ε, πνεύμονα αν θέλετε του, του, του πλανήτη ε, την περιοχή εκεί του Αμαζονίου οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πράγματι η, ε, το σχετικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη ε, εφαρμόζεται ε, στα συνέπεια και τα σχετικά benchmarks ε, θα πρέπει να τηρούνται. Επίσης η Σάντρα Καλίνα ανέφερε στο πλαίσιο της ο, ομάδας παρακολούθησης ότι ασχέτως του πόσο δύσκολες θα είναι διαπραγματεύσεις ενώσο είναι αρμόδια θα συνεχίσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και ε, σε αυτό το πλαίσιο θα καταστήσει σαφές ότι από την πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την υπονόμευση των ε, στόχων όπως αυτοί έχουν τεθεί στο πλαίσιο της συμφωνία των Παρισίων αλλά και ε, παραβιώσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιών δικαιωμάτων, ειδικότερα δε των δικαιωμάτων των αυτόχρονων πληθυσμών. Εάν τελικά καταλήξουμε στην σύνεψη μιας τέτοιας συμφωνίας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ που ζήτησε από τον Herbert να μιλήσει. Ελπίζω όχι πολύ γρήγορα, διότι μιλώντα γρήγορα δυσκολεύεται η δουλειά του διαμηνέων και μόνο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Νομίζω ότι το ζήτημα του Μερκοσούρ πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Αν η συνθήκη τεθεί σε ισχύ, θα αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σόγιας στην Ευρώπη. και θα περιλαμβάνεται κατ' εξουσιοδότηση πράξη για ευνοϊκότερη αντιμετώπιση της σόγιας κατά πάσα πιθανότητα. Η ερώτησή μου είναι τι συνέπειες θα έχει η αυξημένη εισαγωγή σόγιας στην Ευρώπη στην ε, μείωση της δασικής επιφάνειας στην, Αμαζον, στην περιοχή του Αμαζονίου. Αν υπάρξουν μείζονες ε, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την ε, συνθήκη αυτή, από τη συμφωνία αυτή, θα πρέπει με τον αβ τρόπο να τις περιορίσουμε. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να καταστήσουμε τη συμφωνία αυτή περισσότερο δεσμευτική και να μην παραμείνει σε επίπεδο δηλωτικό μόνο. Να δούμε δηλαδή και τις άλλες επιπτώσεις της συμφωνίας. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή. Στην συμφωνία με το Μερκοσούρι η Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει το θέμα της ε, εξαφάνισης του δάσους του Αμαζονίου. Έχετε δει τις τελευταίες εκθέσεις του IPCC όπου γίνεται λόγος για, την περιοχή, για την, τον περιορισμό της χρήσης ε, ζωικών πρωτεϊνών ε, για την τροφή. Εμείς αυξάνουμε την παραγωγή σόγιας για να τρέφουμε τα ζώα. Μήπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορική πολιτική για να μειώσουμε τις ζωοτροφές και κατά συνέπεια την κατανάλωση ζώων. Εγώ έθεσα μια πολύ σαφή ερώτηση. Δεν έχουμε κανέναν εμπειρογνώμονα από την Επιτροπή. Ίσως ωστόσο μπορείτε να μεταφέρετε την ερώτηση και να απαντηθεί στην κυρία Χάουταλα αργότερα. Επόμενο θέμα, ομάδα παρακολούθησης της ομάδας των άνδρων. Έγινε στις 5 Φεβρουαρίου με τον Ματίας Γιώργιανσεν, επικεφαλής ε, της ε, ομάδας για την συμφωνία με την Κολομβία, το Περού και το Εκουαδόρ. με παρουσία και της ε, Προέδρου της ε, Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας του ΝΤΑΓ. Το λόγο σου, κ. Είχαμε ε, κάνει μια πολύ ζωηρή συζήτηση σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, αν θέλετε, της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ε, Περού, Κολομβίας και ε, στο πλαίσιο της προσχώρησης αυτή τη συμφωνία και του σημερινού του Εκουαδόρ ο Σαντιάγο Φίσας και εγώ ήμασταν ε, εκείνοι που προεδρέσαμε στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης ο συνάδελφο είναι αρμόδιο για το Περού και το και εγώ για το Εκουαδόρ που προτίθεται να προσχωρήσει. το Δεκέμβριο έλαβε η τελευταία ε, συνάντηση της Επιτροπής Εμπορικής ε, Πολιτικής ε, στο Κίτο και ο Μάρτιν Γιόργενσον ενημερώθηκε εκεί και πραγματικά είχε μια θετική εντύπωση γιατί όλοι είναι ικανοποιημένοι με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας μέχρι στιγμής και οι συμμετέχοντες από την Κολομβία και από το Εκουαδόρ ε, ήδη θεωρούν ότι με βάση δηλαδή την σύναψη αυτής της συμφωνίας ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ήδη έχει αυξηθεί. Παρ' όλα αυτά, συζητήθηκε το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αύξηση αυτή των, ε, των εμπορικών συναλλαγών και στο μέλλον. Και ζητήθηκε δηλαδή εδώ ε, και άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή πώς ε, οι εμπορικές ροές, η διαφοροποίηση της παραγωγής αλλά και η διασφάλιση των, θέσεων εργασίας και η μείωση των επισφαλών θέσεων εργασία μπορούν να, να, να, να επιτευχθούν. Από εκεί και μετά προβήκαμε σε μια ανταλλαγή απόψεων με την εκπρόσωπο του EU Domestic Advisory Group, της ε, συμβατική δηλαδή ομάδας από πλευρά της Ευρωπαϊκής η οποία συναντήθηκε με ε, τις, ε, όλες τις αντίστοιχες Domestic Advisory ε, Groups εκεί ε, στο Κίτο των υπολείπων χωρών και όπου συζητήθηκε δηλαδή σε βάθος η κατάσταση όπως αυτή ισχύει στις τρίτες χώρες. Άρα λοιπόν η ε, ανάληψη της δράσης και συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτών των τριών domestic advisory groups αξιολογείται ως κάτι το θετικό και έγινε ε, η συζήτηση σε ό,τι αφορά την διεύρυνση αν θέλετε, της δραστηριότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ε, παραδοσιακά ε, στις ε, διάφορες συνάψεις συλλογικών συμβάσεων εργασιών και ούτω καθεξής μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. υπάρχει μια συνδικαλιστική οργάνωση που έχει οριζόντιο διατομιακό χαρακτήρα και έχει καταφέρει να ιδρυωθεί, αλλά η οποία δεν έχει ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αυτής της ε, δομής της εταιρικής ε, σχέσης η οποία έχει ε, δημιουργηθεί ε, στο πλαίσιο των Domestic Advisory Groups. Ε, αυτό δεν ίσχυσε δηλαδή για, την, για τις δύο προηγούμενες χώρες, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε να επιτευχθεί σε σχέση με το Εκουαδόρ. Επίσης, και με την Κολομβία το ζήτημα της καλλιέργειας κόκκας το, οποίο παραμένει ένα πρόβλημα. και εμείς από δική μας πλευρά προτείναμε να υπάρχει μια δυνατότητα επικοινωνία στο πλαίσιο της ε, Domestic Advisory Group με δύο-τρεις ε, προσώπους και θα θέλαμε σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή να βοηθήσει στην διοργάνωση αυτών των ε, και να υποστηρίξει την διοργάνωση αυτών των συναντήσεων σε επίπεδο δηλαδή οριζόντιων ε, ε, ε, επιτροπών έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία, καλύτερη συνεννόηση και καλύτερη εφαρμογή της συμφωνίας. Άρα λοιπόν η εν λόγω συνάντηση της Monitoring Group ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Και ελπίζουμε πως ε, στο πλαίσιο της σύνθεσης του νέου πλέον ε, κοινοβουλίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ κοινοβουλίου και επιτροπής, ε, θα είναι δυνατό να υποστηρίξουμε και να ενισχύσουμε περισσότερο ακόμα τις εργασίες της Domestic Advisory Group σε σχέση με αυτή τη συμφωνία με Κολομβία, Περού και Εκουαδόρ. Επίσης αναφέρθηκε ότι η Βολιβία εξετάζει το ενδεχόμενο σύναψη στενότερων εμπορικών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ότι ενδεχομένω θα ξεκινήσουν ε, συναντήσει έτσι για να βολιδοσκοπηθεί λίγο αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, Δεν βλέπω να ζητάει κανεί άλλο ε, το λόγο, οπότε επανέρχομαι στο ζήτημα τη Μερκοσούπ. Κύριε Σαραφράγκα, συζητήσαμε αυτό το ζήτημα προηγουμένω πριν από τι συνάντηση, γιατί είχαμε προχωρήσει λίγο σύστημα με το χρονοδιάγραμμα, αλλά ενδεχομένω να θέλετε να σχολιάσετε κάτι παραπάνω, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα. Ξέρω ότι αναφέρθηκε ο κύριος Σόλτς το θέμα αυτό. Είχαμε μια συνάντηση της ε, ομάδας παρακολούθησης που έδειξε σαφώς ότι ο τελευταίος γύρος των διαπραγματεύσεων υπό την Προεδρία της Ουρουάης από πλευράς Μπερκοσού δεν έδειξε πρόοδο. Δύο χρόνια, τέσσερα θέματα γυρίζουμε γύρω-γύρω. Αυτοκίνητα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, γεωγραφικές ενδείξεις και θαλάσσιες μεταφορές. Η Προεδρία του Μερκοσούρ πέρασε την 1η Ιανουαρίου στην Αργεντινή που έδειξε καλή διάθεση συνεργασίας για τις διαπραγματεύσεις και από ό,τι μας είπαν ε, στην Επιτροπή βρισκόμαστε σε μια στιγμή διαμόρφωση της θέση της Βραζιλίας κατά βάση λόγω της εκλογής του νέου Προέδρου μπορεί να αλλάξει Υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις στη σχέση μεταξύ Αργεντινής Βραζιλίας. Ο Μπολσονα... Ε, συνήθως ο πρόεδρος της Βραζιλίας όταν ξεκινάει πηγαίνει πρώτη επίσκεψη στην Αργεντινή. Δεν το έκανε ο κ. Μπολσονάρο, πήγε στη Χιλή. Τέλο πάντων, μετά τις αρχικές ε, παρεξηγήσεις ε, μίλησαν μεταξύ τους οι δύο πρόεδροι. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δεσμεύτηκε υπέρ της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσταση ελεύθερου εμπορίου. Αυτή είναι η κατάσταση εν ώψη της επόμενης, ε, ε, του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων το Μάρτιο. Ξέρουμε ότι η πολιτική στιγμή είναι δύσκολη συγκυρία. Είναι δύσκολο να κινητοποιηθεί πολιτικό κεφάλαιο για να λυθεί ε, μια σειρά διαπραγματεύσεων σύμφωνα με την επικεφαλής ε, της, ε, των διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή θα, χρειαστεί, σε, θα χρειαζόταν μια εβδομάδα για να λυθούν τα ζητήματα που μας απασχολούν δύο χρόνια. 30 Απριλίου θα υπάρξει μια συνάντηση της Βρυξέλλες, επίσκεψη Βρυξέλλες από πλευράς του Πρόεδρου της Αρχεντινής. Θα πάει και στη Γαλλία μετά να δει τον Μακρόν. η Επιτροπή, η κυρία με έχει πολιτική βούληση να κλείσει το θέμα στην θητεία τη. Γίνονται διάφορες ε, συναντήσει. Γνωρίζουμε όμω ότι ο χρόνος φεύγει. Στη φάση αυτή η κατάσταση, το ενδιαφέρον και η στρατηγική συμβολή αυτής της συμφωνίας απαιτούν να υπάρξει μια προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Ξέρουμε ότι πολιτικά η συμφωνία αυτή έχει κλείσει κατά 100% πολιτικά, κατά 10% μόνο εμπορικά, μένει εκρεμές ένα 90% των, ε, των εμπορικών ζητημάτων. Είναι δύσκολο, αλλά θα γίνει προσπάθεια τις επόμενες εβδομάδες να προσπαθήσουν να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και μπορούμε να περάσουμε και στη συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης όσον αφορά την Αυστραλία. Η ομάδα παρακολούθησης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εμπορίου και Τουρισμού της Αυστραλίας. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων και μπορεί να μας ενημερώσει ο κύριος Μόιζα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως ήταν μια ανεπίσημη συνεδρίαση και στις 29 Ιανουαρίου επίσης είχαμε και ένα εργαστήριο όσον αφορά τις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Θα θυμούνται οι συνάδελφοι ότι είχαμε δύο γύρους διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και στην ομάδα εργασία ή την ομάδα παρακολούθηση, αν θέλετε, και το εργαστήριο, προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλα τα ευαίσθητα ζητήματα των διαπραγματεύσεων και βέβαια όσον αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τις γεωγραφικές ενδείξεις, την πρόσβαση στην αγορά, τις δημόσιες συμβάσεις, επίσης σε υποεθνικό επίπεδο, υπο-ομοσπονδιακό επίπεδο, ε, στο επίπεδο κάτω από την κοινοπολιτεία δηλαδή. Μας ενδιαφέρουν επίσης οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να εξαχθούν προς την Αυστραλία. Μας ενδιαφέρει εκεί ιδιαίτερα να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιες υπηρεσίες γεωγραφικού εντοπισμού, κάποιες υπηρεσίες ε, δικηγορικές, ε, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες. Εκεί πέρα είναι δύσκολη η πρόσβαση στην αυστραλιακή αγορά. Τώρα από την αυστραλιανή τώρα πλευρά έχουμε τα συμφέροντα όσον αφορά το βοδινό κρέας ε, ή το κρέας από εγωπρόβατα. Στα σημεία αυτά ενδεχομένω οι διαπραγματεύσει είναι δύσκολε. Στο θέμα να βρεθούν βέβαια λύσει. Και θα έλεγα ότι υπάρχει πλέον μια πολύ καλή βάση που μα επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι όντω μπορεί να έχουμε ε, επιτυχεί διαπραγματεύσει ε, ε, προ τα μέσα το τέλο του επόμενου έτου, αν όλα κινηθούν θετικά. Οι εκλογικοί, εκλογικές εκλογικέ διαδικασίε στην Αυστραλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είπαν και οι δύο πλευρέ ότι δεν πρόκειται να επηρεάσουν αρνητικά το χρονοδιάγραμμα. Βέβαια, θα πρέπει τα ευαίσθητα ζητήματα από τεχνική και πολιτική πλευρά να αντιμετωπιστούν μετά τι εκλογέ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι θετικό να λαμβάνονται αποφάσει από του νεοεκλεγεί, θέλετε, τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από την πλευρά της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Μας απασχόλησε το ζήτημα των προτύπων και θεωρήσαμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να επιλύσουμε και άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως για παράδειγμα οι θετικές διατάξεις και τα πρότυπα τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή οι Αυστραλοί στη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ, τα οποία προκαλούν πρόβλημα σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρόσβαση στην αγορά ε, χείριου κρέατος ε, στην Αυστραλία, όπου θεωρούμε ότι υπάρχουν εδώ διάφορα μέτρα υγειονομικής ή φυτονομικής προστασίας που χρησιμοποιούνται κάπως άδικα κατά τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιορίζοντας την πρόσβαση των δικών μας των παραγωγών. Θεωρώ λοιπόν ότι στο πλαίσιο τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα καταφέρουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα ζητήματα ω δέσμη. και αν λάβει η χώρα βέβαια και το Brexit θα πρέπει και αυτό να καλυφθεί στο πλαίσιο τη συζήτηση που γίνεται για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Αυτά είχα να σα πω. Πολύ ωραία. Υπάρχουν παρατηρήσει. Δεν βλέπω κανένα, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε έτσι και το σημείο 6 τη ημερήσια διάταξη. και θα κάνουμε ένα διάλειμμα 14 λεπτών έτσι ώστε να ξεκινήσουμε στις 10 ακριβώς ε, τις ψηφοφορίες μας. Okay. Ladies and... Uh, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ πολύ. We will start quite soon with our... Θα αρχίσουμε σύντομα με τις ε, ψηφοφορίες μας. Good. Πολύ ωραία. Προτού ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία όμως, θα ήθελα να καλωσορίσω ορισμένα μέλη από την μια Επιτροπή Παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν τις εργασίες της δικής μας Επιτροπής από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ας κάνουμε μια δοκιμή, δοκιμαστική μάλλον ψηφοφορία, να δούμε αν λειτουργούν οι συσκευέ, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Τέλεια, όλα τέλεια. Πρώτη ψηφοφορία, εφαρμογή του κανονισμού GSP, συμβαστική Παρεθμόν 1 πέρα παρακαλώ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 121 μια πρόταση έχουμε εδώ επιπλέον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 106 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά,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 εγκρίνεται. 35 και 36 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση για τις τροπολογίες 35 και 36 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 39 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 39 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 41, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση και τροπολογία 43, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται σαφώς. 44 τώρα υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 49. Άρτη ψηφοφορία. Πέρασε εγκρίνεται. 49 υπέρ. Σα το συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, την ψηφίσαμε αυτήν. Συμβασική τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας το ελέγξουμε. Άρτη ηλεκτρονική ψηφοφορία για τροπολογία 59. Πέρας. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. άρθρη ψηφοφορία παρακαλώ για την τροπολογία 2. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12, 13 και 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 15 και 16 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 17, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 21 και 22 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24-25 μαζί ήταν ταυτόσιμες. 26 με προφορική τροπολογία υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος η τροπολογία 27 άρτη ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται η γνωμοδότηση τώρα από την ΑΦΕΤ εκτιμώντας ΣΥΠΕΡ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Και απορρίπτεται. Περνάμε στο λογική σκέψη D υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τολική σκέψη D, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 19 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρτη ψηφοφορία, παρακαλώ, για την παράγραφο 19. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παράγραφο 20. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη γνωμοδότηση Επιτροπής Ανάπτυξης τώρα. Όχι, σας ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Έχουμε και την παράγραφο 22 να ψηφίσουμε. Παράγραφο 22, λοιπόν. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα περνάμε στη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΔΕΒΕ, παράγραφος 3, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 13, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Και μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται η έκθεση. Next item is item 8. Επόμενο θέμα, 8. Σύσταση για την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ένωσης και ΕΠΑ. Συμβιβαστική 6 πρώτα πρώτα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Α. Υπέρ Συγγνώμη, τη 48, τροπολογία 48. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7α υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 61 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα κάνουμε έναν έλεγχο για την 61, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται.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 Απορρίπτεται νομίζω, αλλά το ξαναβλέπουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9α υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 9α. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 71, μία πρόταση, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για την 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά, αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 10α υπέρ, κατά, άποχες, έλεγχος. Για την 10α άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 81, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10β υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για τη 10β. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά στο δούμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11α υπέρ. Κατά. Είναι ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζουμε να ψηφίζουμε λοιπόν. 11A, the vote is open. 12α. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 93. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ονομαστική ψηφοφορία για την συμβιβαστική 12α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος για την 24 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 σε 2 τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 και 36 μαζί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ή ηλεκτρονικός έλεγχος για την 35 και 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο Vote is Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ 17 κατά. Point Σημείο 9. Παρακαλώ. Χάιντι. Ευχαριστώ, πρόεδρε να σας ενημερώσω ότι ήθελα να εφαρμόσω το νέο κανόνα, το νέο άρθρο 11.3 για τα, τις υποχρεώσεις των εισηγητών να συμπεριλάβουν ένα κατάλογο των ατόμων και φορέων ε, των οποίων ακούσαμε την άποψη. Είναι μια μεγάλη, ένας μεγάλος κατάλογος και ελπίζω να συμπεριληφθεί στο κείμενο που θα πάει στην Ολομέλεια, διότι έχει τους πάντες από τον Πρωθυπουργό του Βιετνάμ, και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Βιετνάμ μέχρι τις μεγάλες ΜΚΟ, καθώς και δύο πρέσβεις χωρών της Ένωσης. Ελπίζω να αποτελέσει πηγή έμπνευση για τους υπόλοιπους από εσάς, όταν ετοιμάζετε νέες εκθέσεις. Ευχαριστώ, όπως ξέρετε, γκρίναμε τους νέους, ε, το νέο εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου με τις απαιτήσει αυτές για εισηγητές προέδρους να ενημερώνουν τα μέλη με ποιους έχουν συζητήσει. Προς το παρόν το προσωπικό του Κοινοβουλίου εργάζεται ώστε να διαμορφώσει μια πλατφόρμα στο ίντερνετ που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους με ευκολότερο τρόπο από ό,τι εσείς στη δουλειά σας. Τροπολογία 2. Συμβαστική 2 εννοεί. Υπέρ αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω, το ελέγχουμε για την 2α άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται προφανώς συμβιβαστική 2β υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2γ 2σ υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 λέει ο πρόεδρος κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5α υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5β υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, μία υπέρ κατά αποχές δεκτή, δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γνωμοδοτής επιτροπών. Δεύε. Δεύε τρία υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΔΕΒΕΠΤΑ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η ηλεκτρονική πληροφορία για το τελικό κείμενο άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Μία αποχή μόνο, όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Συγχαρητήρια. Σημείο 10. Σύμφωνη γνώμη για την συμφωνία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Δεκτή η σύμφωνη γνώμη. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Αποφασίσαμε στο ξεκίνημα της συνεδρίασής μας να αναβάλουμε το σημείο 11. Πάμε λοιπόν στο σημείο 12. Αν θέλετε τώρα να φύγετε, παρακαλώ να φύγετε προσεκτικά και χωρίς φασαρία. Θα κάνω διάλειμμα πάντως για ένα λεπτό για να φύγετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 12 της μερίσιας διάταξης. Στις περισσότερες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών έχουμε ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την εξαίρεση βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά όμως, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να εξετάζουμε τα όσα περιέχονται σε αυτό το κεφάλαιο εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης και μια σημαντική πτυχή στο κεφάλαιο αυτό είναι ο ρόλος που δραματίζουν οι εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες. Οι βασικοί εκπρόσωποι σε αυτές τις εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες στο πλαίσιο τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Όσον αφορά λοιπόν τα καθήκοντά τους, αρμοδιότητές τους, αλλά και την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 137 του κανονισμού, τους ζητήσαμε να υποβάλουν γνωμοδότηση όσον αφορά την λειτουργία αυτών των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, Μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Αλμπέρτο Μάτσολα, ο οποίος είναι ο, ο εισηγητής εκ μέρους Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό και έχει στη θέση του 7 λεπτά για να μας παρουσιάσει την γνωμοδότησή του. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστούμε για αυτό το αίτημα προς ε, την ε, ό,τι σε ό,τι αφορά τη σύνταξη γνωμοδότηση, ό,τι αφορά αυτές τις εγχώρες συμβουλευτικές ομάδες. Και αν μου επιτρέπετε θα συνεχίσω στα Ιταλικά. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή στι 11 Οκτωβρίου έλαβε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την σύνταξη γνωμοδότηση όσον αφορά τι εσωτερικέ συμβουλευτικέ ομάδε και όσον αφορά την επέκταση των αρμοδιοτήτων και την καλύτερη λειτουργία των ομάδων αυτών. Τρει ομάδε μελέτη διοργανώθηκαν, δύο συνεδριάσει του τμήματο του δικευμένου, όπου είχαμε έντονε συζητήσει και είχαμε και ψηφοφορίε στην ολομέλειά μα όπου είχαμε εκεί και κάποιες τελικές τροπολογίες όπου πέρασε μια διαφορά 80-70 ψήφων. Εν τέλει εγκρίθηκε η γνωμοδότηση αυτό, αυτή με 150 ψήφους υπέρ και δύο αποχές. Θα έλεγα λοιπόν ότι συμμερίζονται οι περισσότεροι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τη γνωμοδότηση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το εμπόριο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, Αναγνωρίζουμε όμως επίσης ότι ε, υπάρχουν ε, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία δεν κατανέμονται ισότιμα σε όλα τα κράτη-μέλη και σε όλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Η ΣΕΤΑ, η Συμφωνία TTIP κατέδειξαν θεωρώ πραγματικά ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ένταση και ενδιαφέρον όμως από τους πολίτες όσον αφορά την έγκριση των συμφωνιών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών σε όλε αυτέ τι συμφωνίε. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ θεσμικών οργάνων και κυβερνήσεων δεν μπορούν να αποτελούν τη μόνη πτυχή των συμφωνιών αυτών. Κατά την άποψη λοιπόν της ΕΟΚΕ, οι εσωτερικές αυτές συμβουλευτικές ομάδες θα πρέπει να έχουν έναν ρόλο, ο οποίο να μην είναι μόνο εκτελεστικός, αλλά και γνωμοδοτικός και συμβουλευτικό και θεωρούμε ότι θα πρέπει οι ομάδες αυτές να θεσμοθετηθούν, να επισημοποιηθούν στα πλαίσια των συμφωνιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλύπτουν όλες τις πτυχές των συμφωνιών και να εκπροσωπούν ισότιμα και τις τρεις ομάδες που έχουμε στην ΕΟΚΕ, δηλαδή εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των λοιπών συμφερόντων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι ομάδες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές που έχουν να κάνουν με την απασχόληση, να αναφέρονται επίση στι συμβάσει τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία, να αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, στι περιβαλλοντικέ επιπτώσει, στα συμφέροντα των καταναλωτών, καθώ επίση και στι υπόλοιπε πτυχέ τη οικονομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει όλες οι πτυχέ των εμπορικών συμφωνιών μα να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασία από τι εσωτερικέ συμβουλευτικέ ομάδε. Αυτή τη στιγμή καλύπτουμε κυρίω μόνο την πτυχή που έχει να κάνει με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σαφώ θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή των ομάδων αυτών σε όλε τι πτυχέ των συμφωνιών. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο και οι χώρε εταίροι θα καταφέρουν να αποδεχτούν πολύ πιο εύκολα την παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών Υπάρχουν πολλέ κυβερνήσει ή χώρε εταίρειε που δεν το αποδέχονται εύκολα ακόμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια κοινή ομάδα ε, συμβουλευτική που να εκπροσωπείται η κοινωνία των πολιτών τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις ε, χώρες εταίρους. Ξέρετε ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή μια κοινή ομάδα, όπω για παράδειγμα έχουμε ήδη στη συμφωνία με τη Χίλη. Δεν υπάρχει λόγο να δημιουργήσουμε νέε συμβουλευτικέ ομάδε, Όσον αφορά τη σύνθεση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο μηχανισμό επιλογή των μελών των ε, εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων και εμεί ω ΕΟΚΕ μπορούμε να συμβάλλουμε στην καλύτερη αυτή δυνατή επιλογή όσον αφορά την ε, λειτουργία, την ε, οργάνωση των εσωτερικών συμβολευτικών ομάδων θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις ετησίω. Πολύ συχνά τώρα γίνεται μόνο μία. Στην ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να έχουμε δύο συνεδριάσεις μεταξύ ευρωπαϊκής πλευράς και της πλευράς εκείνης από την χώρα εταίρο και θα πρέπει βέβαια να γίνεται τουλάχιστον μια συνεδρία ετησίω ενώπιο, εν οποίο οι υπόλοιπε μπορούν να γίνουν μέσω τηλεδιασκέψεων αλλά να προβλέπετε τουλάχιστον μία συνεδρίαση που θα γίνεται με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κάθε χρόνο διάσκεψη όλων των μελών των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων, προκειμένου να καταστεί δυνατή αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών από τι αντίστοιχε ομάδε και θα πρέπει επίση να έχουμε την ε, δυνατότητα να ακούμε και να διαβουλευόμαστε μέσω μιας αιτήσιας ακρόασης και με άλλους ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Καθώ επίση και με άλλε ομάδε που έχουμε σε διάφορες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να ευρύνουμε λίγο την αρμοδιότητά μα. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε όλε τι προτεραιότητε που θα πρέπει να έχουμε, Πάντω, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να καλύπτουμε όλε τι πτυχέ των συμφωνιών, όπω σα είπα. Μία άλλη πρόταση που κάνουμε. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτέ οι εσωτερικέ συμβουλευτικέ ομάδε να υποβάλουν τι δικέ του συστάσει και έπειτα ο Πρόεδρός του θα πρέπει να μπορεί να τις υποβάλει και στα πλαίσια της Επιτροπής για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να μπορούμε να λαμβάνουμε και κάποιες απαντήσεις, μια, κάποια ανταπόκριση αν θέλετε, στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου και Βιώσιμης Ανάπτυξης όσον αφορά τις προτάσεις μας αυτές. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή προτού συσταθούν αυτές οι έσω, ξεκινά με κάποιες διαπραγματεύσεις και άλλες δραστηριότητες με τις χώρες εταίρους. Αυτό είχαμε κάνει και με την Ιαπωνία. Προτού συσταθεί η επίσημη ε, εσωτερική συμβουλευτική ομάδα με την Ιαπωνία, είχαμε ήδη έρθει σε διερευνητικέ επαφέ με τη χώρα αυτή. Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει είναι η χρηματοδότηση, ιδίω στι τρίτε χώρε. Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μα. Θεωρούμε λοιπόν ότι στο κείμενο των συμφωνιών θα πρέπει να βλέπονται συγκεκριμένε ρήτρε για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων, ιδίω από τι χώρε εταίρου. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή θέλει να έχει συνεχή παρουσία στο πλαίσιο των ομάδων αυτών. Βέβαια, θα πρέπει εδώ πέρα να πούμε ότι ο αριθμός των συμφωνιών αυξάνεται όλο και περισσότερο. Επομένω, θα δυσχεράνει και το δικό μας το έργο και από χρηματοδοτική πλευράς. Τα επόμενα πέντε χρόνια, τα επόμενα τρία μάλλον χρόνια, αναμένεται να διπλασιαστεί το κόστος της παρουσίας της ΕΟΚΕΣ τη ΕΣΟ και θα τριπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να συμμετέχουν 77 μέλη σύντομα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στι διάφορε εσωτερικέ συμβουλευτικέ ομάδε. Θα πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να αυξήσουμε την χρηματοδότηση για τι ομάδε αυτέ και θα πρέπει η χρηματοδότηση αυτή να αντικατοπτρίζεται πραγματικά στο προπολογισμό που μας επιτρέπει να έχουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα δύο ακόμα τελευταίες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω δεν ε, είναι απαραίτητο να έχουμε και με τις 69 χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες, πρέπει να έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια για τη θέσπιση των έσω αυτό και τον καθορισμό του αρισμού των μελών. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι όγκος του εξωτερικού εμπορίου, οι εμπεδίσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα της χώρας εταίρου, η σημασία της συμφωνίας από γεωπολιτική και στρατηγικής άποψης, καθώς και οι σχετικές με τη βιωσιμότητα πτυχές. Οι έσω αυτές ε, θα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μπορούν να ε, υποβάλουν, να υπάρχουν μάλλον οι αυτές, κάθε φορά που έχουμε επενδύσει που υπερβαίνουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ως ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή θα θέλουμε να μπορούμε να υποβάλουμε εκθέσεις όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και αυτά είναι τα βασικά σημεία της γνωμοδότησής μας. Ευχαριστώ. Yeah. Σας ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. είναι πρώτη. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρώ πως ε, πρόκειται εδώ για μια εξαιρετική πρόταση από την πλευρά της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ε, ε, το να περιλαμβάνεται δηλαδή περισσότερη κοινωνία των ε, πολιτών στην υλοποίηση αυτών των συμφωνιών ελευθερίου εμπορίου. Ε, και εμεί ε, πραγματικά συμφωνώ στο να υιοθετηθεί αυτή η πρόταση από την πλευρά τη Επιτροπή και του Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα να θέσω και κάποια ερωτήματα. Καταρχήν, η ΕΟΚΕ θεωρεί πω για το κεφάλαιο τη βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να ισχύουν και κυρώσει. Και αν ναι, εάν προβλέπεται ένα τέτοιο μηχανισμό κυρώσεων, η ΕΟΚΕ θεωρεί πως θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο εδώ, να παίζουν οι εγχώριες συμβουλευτικές ομάδες. Ένα ακόμα ερώτημα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθοράς, για παράδειγμα, στο πλαίσιο συμφωνιών όπω Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Χιλή, θα πρέπει να παίζουν κάποιο ρόλο αυτέ οι χώρε συμβουλευτικέ ομάδε. Ε? Ε, και σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και πάλι θα πρέπει να παίξουν κάποιο ρόλο. Για παράδειγμα, στην ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Μεξικού. Ε, Πώ μπορούν να παίξουν έναν ενεργό ρόλο σε αυτά τα επίπεδα οι ε, χώρε συμβουλευτικέ ομάδε. Ε, και ένα τέταρτο και τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξή. Στο 1-3 τη γνωμοδότησή του, της, η ΕΟΚΕ θεωρεί πως ε, τα συμφέροντα του συνόλου της ε, κοινωνίας θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο πλαίσιο ενός κοινού φόρουμ. Ε, για να το επιτύχουμε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην λάβει ακριβώς έναν κλειστό, αν θέλετε, χαρακτήρα περιχαρακωμένο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Η Μαρία Αρένα έχει το λόγο. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής για την έκθεση Ευρωπαϊκής Οικονομικής ε, Επιτροπή, έχω τρεις ερωτήσει. Πρώτον, για την ε, προσέγγιση του στο θέμα των κυρώσεων, το ΙΟΚΕ θέλει το Domestic Advisory Group να δουλεύει για το σύνολο της έκθεσης. Έχει εξετάσει το θέμα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν καλύπτεται από το θέμα της διαχείρισης του Dispute Settlement System. Ε, μπερδεύομαι αγγλογαλικά. Το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη δεν καλύπτει από αυτό το μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Μήπως θα έπρεπε να διευρυνθεί αυτό σε, όλες τις, ε, σε όλη τη συμφωνία. Τρίτη ερώτηση. Τι, γίνονται με τις, τι γίνεται με τις συστάσεις, είναι απλώς γνωμοδοτήσεις ή πρέπει να ενσωματώνονται υποχρεωτικά και στην ενεργοποίηση των ρητών διασφάλισης, για παράδειγμα, αν ε, εμφανίζεται ότι μία σύσταση που διατυπώθηκε θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα διασφάλισης της εμπλεκόμενης χώρας, θα ήταν ενδιαφέρον. Και τι γίνεται με την ενεργοποίηση αυτών των συστάσεων στις ρήτρες αναθεωρήσεις που ζητούν πλέον μόνιμα οι εμπορικές συμφωνίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Κίρτον Αναγκάλη, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για αυτή την έκθεση, την ομοδότηση. Και εγώ θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα και να κάνω κάποια σχόλια. Ε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό που ακούστηκε ότι δεν ε, χρειάζεται απαραίτητο να υπάρχει μια εγχώρια συμβουλευτική ομάδα για όλες τις συμφωνίες, ε, θα ήθελα ε, να πω πως είναι κάπω προβληματικό γιατί εάν πραγματικά είναι ζήτημα προτεραιότητα ε, αυτό του εμπορίου και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ε, ε, τότε θα ήταν προβληματικό το να λέμε ότι σε κάποιε περιπτώσει χρειαζόμαστε ναι, απαραίτητο κάποιε εγχώριε συμβουλευτικέ ομάδε, αλλά σε κάποιε άλλε περιπτώσει, σε άλλε συμφωνίε όχι. Δηλαδή, ποιο θα ήταν αρμόδιο για να αποφασίζει ότι έχουμε ένα πρόβλημα, αν θέλετε, σε σχέση με κάποια χώρα. ειδικότερα στο πλαίσιο δηλαδή ε, ε, ε, μεγάλων, μεγάλου όγκου, αν θέλετε, συμφωνιών που καλύπτουν δηλαδή πολύ σημαντικά μπλοκ, Ενδεχομένως, αν δεν υπάρχει σε συμβουλευτική ομάδα, να μην λάβουν την κατάλληλη σημασία τα ζητήματα που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα μενοτήτων και ούτω καθεξής. Κάτι ακόμα τώρα πολύ σωστά αναφέρει η δική σα νομοδότηση τη μεγάλη πρόκληση και το μεγάλο πρόβλημα που αποτελεί ε, η έλλειψη των πόρων. Δηλαδή, αν θέλουμε πραγματικά να θέσουμε στον καρδιά των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου τη βιώσιμη ανάπτυξη, τότε θα πρέπει να διαθέσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Και θα πρέπει να παράσουμε και την κατάλληλη υποστήριξη έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα όσα συμβαίνουν μέσα στι εγχώριε συμβουλευτικέ ομάδε έχουν πραγματικό αντίκτυπο στι ε, εκάστοτε εμπορικέ σχέσει. Ε, η ιδέα του ο πρόεδρος της εκάστοτε ε, συμβουλευτικής ομάδας να λογοδοτεί στην αρμόδια εμπορική επιτροπή πράγματι θα μπορούσε να διασφαλίσει αυτή την άμεση σχέση. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις νέες διαδικασίες υποβολή παραπάνω των προσφυγών τι σκέφτεται η ΟΚΕ, δηλαδή σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στις ε, εν λόγω συμφωνίες. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τέτοιου είδου διαδικασίε υποβολή παραπάνω σε ό,τι αφορά παραβιάσει, για παράδειγμα, εργασιακών δικαιωμάτων, παραβιάσει κανόνων σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική προστασία και ούτω καθεξής. Ε, θεωρούν ότι θα μπορούσε, θεωρεί ότι θα μπορούσε να υπάρχει ένας τέτοιος μηχανισμός ε, ε, υποβολής παραπώνων και θα μπορούσε να λειτουργήσει σε συνάρτηση με το ρόλο των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων. Ένα τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θέσω είναι ότι υπάρχει ανάγκη να διασφαλίσουμε τη συγκέντρωση, αν θέλετε, εμπειρίας από τις συμφωνίες ε, που έχουμε ήδη κάποια χρόνια που ε, τρέχουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε αποκομίσει κάποια εμπειρία από τη λειτουργία ορισμένων ε, χώρων συμβουλευτικών ομάδων, ορισμένες φορές ανετική εμπειρία, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω την ΕΟΚΕ κατά πώς θεωρεί ότι θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να συγκεντρώσουμε όλη αυτή την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Η ανησυχία μου είναι δηλαδή να υπάρξει υπερβολική φθορά αν θέλετε με την αλλαγή των μελών και ούτω καθεξής. Δηλαδή με άλλα λόγια πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα είδος ιστορικού για αυτές τις εγχώριε συμβουλευτικές ομάδες, ένα είδος δηλαδή δόμησης της εμπειρίας τους έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, για παράδειγμα, που έχουμε ε, αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο τη συμφωνία ε, με την ε, Κορέα, όπου δηλαδή εδώ και χρόνια έχουν τεθεί κάποια προβλήματα στο πλαίσιο των χώρων συμβουλευτικών ομάδων, αλλά μόλι τώρα η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση. Άρα λοιπόν, πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια σε ό,τι αφορά τι εργασίε αυτών των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Υπάρχει κάποιο άλλο μέλο που θα ήθελε να πάρει το λόγο. Εάν όχι, θα δώσω φυσικά το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Μαντλέν Τουνίγκα, η οποία είναι αρμόδια για αυτό το ζήτημα των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων. Είναι από την μονάδα της, ε, του εμπορίου και της ε, βιώσιμης ε, ανάπτυξης και θέτω και εγώ το ερώτημα που έθεσαν οι συνάδελφοι, δηλαδή πώς σκοπεύει να εφαρμόσει στην πράξη αυτή την σύσταση από την πλευρά της Οικονομικής και κοινωνική επιτροπή. Καλημέρα σα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για ε, την κατάρτιση αυτή τη ε, ιδιαίτερα περιεκτικής ε, γνωμοδότησης, αυτή της έκθεση. Άλλωστε βρισκόμασταν σε στενή συνεννόηση μαζί της και νομίζω πως μπορείτε να είστε περήφανοι γιατί συγκεντρώνεται εδώ την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από το 11 και μετά. Πραγματικά μπορείτε να είστε ε, περήφανοι για αυτή την έκθεση. Ε, προφανώς ε, εγώ παίρνω το λόγο εδώ, αλλά δεν πρόκειται για αρμοδιότητα μόνο ε, της δικής μου μονάδας. Έχω ε, εξ μου και τον Πίτερ Σάντλερ που ασχολείται με τα θεσμικά ζητήματα και τα ζητήματα κοινωνία των πολιτών. Και βέβαια, όπω γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, στο πλαίσιο τη οποία θα διευρύνουμε ε, τα ζητήματα της, ε, των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και τα στήματα κοινωνίας των πολιτών, καταρχήν σε σχέση με το Μεξικό, Μεξικό και τη Χιλία και στο μέλλον και στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών αυτού του χαρακτήρα, οπότε θα έχουμε περισσότερους συναδέλφους που θα είναι αρμόδιοι, περισσότερες μονάδες. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, να σα αναφέρω τι δράσει τι οποίε έχουμε αναλάβει σε αυτό το τομέα. Καταρχήν, να σα πω πω είμαστε περήφανοι για το γεγονό ότι έχουμε πολλέ ε, ε, συναντήσεις, για παράδειγμα 22 με 25 ετησίως ε, με την ε, κοινωνία των πολιτών, το 1 τρίτο εκ των οποίων συναντήσεων αφορά τις ε, συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Μετά έχουμε τις ομάδες επαφής σε ό,τι αφορά το εμπόριο και στη συνέχεια έχουμε και τις, φωνή, τις ομάδες σε ό,τι αφορά τις την βιώσιμη ανάπτυξη. Έξι φορές συνεδρίωσε, μετά είχαμε τη μεγάλη διάστευση η οποία έλαβε χώρα, αλλά από εκεί και μετά workshops, ε, σεμινάρια. Είχαμε 27 ε, συναντήσεις και στις Βρυξέλλες και αλλού ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τώρα των στόχων της βιώσιμη ανάπτυξης και την υλοποίησή της. Είχαμε πολλές συναντήσεις και με την ΕΟΚΕ και συνδιοργανώσαμε την σχετική διάσκεψη από κοινού τον Επίτροπο και δώσαμε συνέχεια στο σχέδιο δράσης των 15 σημείων. Επίσης έχουμε τακτικές συναντήσεις με τη γραμματέα του τμήματος ε, REX ε, και το ίδιο το τμήμα REX και τις ε, ομάδες μελέτης του από την πλευρά της ΕΟΚΕ και πάντοτε προσπαθούμε εδώ να βρισκόμαστε σε συνεννόηση, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό γιατί ακριβώς ε, παίζει ε, το ρόλο ενός ε, ατύπου συμβουλευτικού σώματος το ΡΕΞ. Από εκεί και μετά έχουμε συναδέλφου με τους οποίους βρισκόμαστε σε επαφή τόσο από την ΕΟΚΕ όσο και από τις εγχώριε συμβουλευτικέ ομάδες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολύ σημαντική βάση για τις περαιτέρω εργασίε μας. Καταρχήν με ρωτήσατε ε, ποια είναι η συνέχεια που θα δώσουμε σε αυτή την ε, νομοδότηση. Καταρχήν υπάρχει μια επίσημη διαδικασία. Ε, δηλαδή, όταν υπάρχει μια νομοδότηση από την ΕΟΚ, εμεί έχουμε τρει μήνε στη διάθεσή μα ε, και βρισκόμαστε ακριβώ στη φάση αυτή τη διαβούλευση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα αναμείνουμε ε, τρει μήνε και θα συνεχίσουμε στο πλαίσιο αυτή τη περίοδου τι ε, άτυπε μα συζητήσει με την ΕΟΚ σε ό,τι αφορά τι συστάσει που κάνει στη γνωμοδότηση. Όπω είπα, κατά την τη παρέμβαση μου, η ΕΟΚΙ έχει πραγματικά ε, κάνει εξαιρετική δουλειά εγώ και ε, πραγματικά εδώ ε, βλέπουμε να με επιτυχία, να στέφεται με επιτυχία αυτή η συμπερίληψη του, του πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών μέσα σε αυτές τις ε, συμφωνίες που το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, μόνος παίκτης παγκοσμίω. Ε, βλέπουμε δηλαδή να είναι αποτελεσματικέ οι διατάξει που έχουμε προβλέψει. Τώρα, κάνετε κάποιε συστάσει οι οποίε είναι πολύ ευπρόσδεκτε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ζήτημα τη επικοινωνία. Ε, Αυτό είναι ο τέταρτο επιλώνα ε, του σχεδίου δράση των 15 σημείων μα, δηλαδή διαφάνεια και επικοινωνία. Κρίσιμη λοιπόν σημασία σε αυτό το σημείο. Αλλά και περαιτέρω σημεία επί των οποίων εργαζόμαστε είναι η διεύρυνση του πεδίου αρμοδιότητα, αν θέλετε, στο πλαίσιο μελλοντικών συμφωνιών, έτσι ώστε όλα τα ζητήματα να καλύπτονται σε ό,τι αφορά το σύνολο της συμφωνίας ε, και άρα θα καλύπτονται και τα σημεία τα οποία αναφέρατε εσείς, ε, για παράδειγμα τα ε, συμφέροντα των καταναλωτών. Από εκεί και μετά. σε ό,τι αφορά τώρα τις υποχρεώσει, ε, τι δεσμεύσει ανάλυση υποχρεώσεων. Προφανώ δεν μπορούμε να το περιλάβουμε μέσα σε αυτόν τον προπολογισμό, αλλά ε, στο πλαίσιο των σχετικών ε, project έχουμε για παράδειγμα προβλέψει τα 3 εκατομμύρια ευρώ ως μέρο του προπολογισμού σε ό,τι αφορά έξοδα ταξιδίου και από εκεί και μετά διοργάνωση και workshops σε ό,τι αφορά τα διάφορα φόρα της κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε ακριβώ να δώσουμε περισσότερη έμφαση. Ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα που αναφέρει η γνωμοδότηση είναι η επιμονή, αν θέλετε, στη βελτίωση αυτών των ε, συμφωνιών και μέσω, για παράδειγμα, της ε, ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών και θα συνεχίσουμε ακριβώς την διοργάνωση των ε, σεμιναρίων. Όλα αυτά, λοιπόν, αναφέρονται μέσα στη γνωμοδότηση. Από εκεί και μετά υπήρξαν ένα-δύο σημεία επί των οποίων δεν είμαστε ε, υποχρεωτικά τη ίδια άποψη με την ΟΚΙΟ, παρότι αντιλαμβανόμαστε τη συλλογιστική τη. Κατά τη δική μα άποψη, οι χώρε συμβουλευτικέ ομάδε θα πρέπει να παραμείνουν ανεξάρτητε και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε κάποιο θεσμικό όργανο προκειμένου να γίνεται από αυτό η επιλογή των μελών ή προκειμένου να, η προεδρία να γίνεται από εκείνο. Δηλαδή, αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να ρυθμίζονται από την ίδια την εγχώρια συμβουλευτική ομάδα. Επίση, θεωρούμε πω αυτέ οι ομάδε θα πρέπει να παραμείνουν όσο το δυνατόν πιο διαφανεί και πιο ανοιχτέ στι ε, ομάδε τη κοινωνία των πολιτών και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να διορίζονται από την κυβέρνηση. Θα πρέπει δηλαδή ε, ακριβώς με έναν ανοιχτό χαρακτήρα να δίνεται ε, περισσότερη ε, σημασία, περισσότερη έμφαση στις μικρότερες ε, κλίμακες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δεν λαμβάνουν υποστήριξη από την κυβέρνηση. Τώρα υπήρξαν κάποια ακόμα ερωτήματα που θέσατε γνωρίζετε την άποψη, για παράδειγμα, της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα όσα σχολιάζεται, σε ό,τι αφορά την επίλυση διαφορών. Όλες οι συμφωνίες περιλαμβάνουν μηχανισμούς δεσμευτικούς επίλυσης διαφορών. Όπως γνωρίζετε, ξεκινήσαμε ε, μια ε, πρώτη διαδικασία με την Κορέα και βρισκόμαστε σε διακυβερνητική διαπραγμάτευση, δηλαδή στα τέλη του Μαρτίου ε, ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία, οπότε μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε αποφασίσει κατά πόσο θα διορίσουμε ένα πάνελ ή όχι. Οπότε πράγματι υπάρχει ένα ε, μηχανισμός επίλυσης διαφορών ο οποίο λειτουργεί στην πράξη και θα πρέπει να δούμε τι θα αποφέρει τελικά. Και βέβαια πρόκειται για την πρώτη φορά που αξιοποιούμε αυτό το μηχανισμό επίλυση διαφορών στο πλαίσιο μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Από εκεί και μετά υπήρξε και ένα ερώτημα περαιτέρω που τέθηκε, το οποίο δεν είμαι βέβαια αν κατάλαβα σωστά, σε ό,τι αφορά τι συστάσει ε, και ε, ρήτρε διασφάλιση, safeguard clauses. Ε, ε, ευχαριστώ σα θα δώσω αργότερα κάποιες απαντήσεις. Μετά, σε ό,τι αφορά ε, τις ρήτρες αναθεώρησης των συμφωνιών, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Καναδά, ε, εργαζόμαστε από αυτού. Θέλουμε δηλαδή στο πλαίσιο μιας τέτοιας αναθεώρησης να αξιοποιήσουμε την εμπορία που θα έχουμε συλλέξει για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη συμφωνία. Τώρα, ε, η πόροι, μάλλον η έλλειψή τους αποτελεί μια πρόκληση για όλους, αλλά εμείς είμαστε 23 άτομα, ως ε, δηλαδή ε, προσωπικό ε, στην δική μου μονάδα και Εξετάζοντα ε, τα ζητήματα τα οποία καλύπτουμε στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, να πω ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με την κατάσταση πριν ένα-δύο χρόνια. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ε, διαδικασία υποβολής παραπώνων ή προσφυγών, όπως αναφέρουμε και στο σχέδιο δράσης, εμεί πράγματι παρακολουθούμε τέτοιου είδους παράπονα, ε, προσφυγέ. Για παράδειγμα έχουμε λάβει ε, ένα τέτοιο παράπονο σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με το Περού και έχει πολύ περίπλοκο χαρακτήρα αυτό το παράπονο, οπότε εμείς ε, σε αυτή τη φάση προετοιμάζουμε μια απάντηση απέναντι σε εκείνου δηλαδή οι οποίοι υπέβαλαν αυτό το παράπονο. Πάντως στο πλαίσιο της όλης της διαδικασίας ήμασταν σε στενή επαφή μαζί τους, μεταβήκαμε και στο Περού για να κάνουμε μία συλλογή εκεί στοιχείων, οπότε θεωρούμε πως ε, ε, δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερο μηχανισμός. Δηλαδή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ε, παράπονα στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων. Αυτά από την πλευρά μου. Βλέπω και τους συναδέλφους, δεν βλέπω ότι να θέλουν να προσθέσουν κάτι, οπότε σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για αυτή την πολύ ουσιαστική νομοδότηση. Ευχαριστώ μία ερώτηση από πλευρά μου για την ρήτρα επανεξέτασης. Και στη ΣΥΤΑ και στην Ιαπωνία το έχουμε. Ξέρετε την άποψη του Κοινοβουλίου. Έχετε τώρα και τη γνωμοδότηση και θέση της ΕΟΚΕ. Okay. Πώς θα ενσωματώσετε αυτές τις γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία ε, επανεξέτασης ε, του κεφαλαίου για την επίλυση των διαφόρων ιδιαίτερα στο Καναδά Έχουμε αυτή την συμφωνία ήδη σε ισχύ εδώ και 1,5 χρόνο. Πώς είναι η κατάσταση στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Ε, η συμφωνία με την Ιαπωνία τώρα μόλις τέθηκε σε ισχύ. Μπορώ να σας πω για τον Καναδά. Ίσως θυμάστε στα κοινά συμπεράσματα, τα κοινά πρακτικά δεν ξέρω πώς τα ονομάζουμε. Δεν στην, στην τελευταία συνάντησή μας ε, που υποβλήθηκε και στην Επιτροπή Εμπορίου, συμφωνήσαμε επί ενό προγράμματος εργασίας. Έχουμε λοιπόν επαφές με τον Καναδά για να συζητήσουμε το περιεχόμενο και την κατεύθυνση αυτή της ρήτρα επανεξέταση και θα υποβάλουμε τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Εμπορίου. Αυτή είναι η δουλειά αυτή τη στιγμή. Μπορεί να πείτε ότι η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ πριν 1,5 χρόνο, αλλά για να γίνει η αναθεώρηση μιας συμφωνίας πρέπει να υπάρξει και μια εμπειρία. Να δούμε τι λειτουργεί και τι όχι και τι πρέπει να κάνουμε. Βρισκόμαστε στη φάση αυτών των συζητήσεων. Είχαμε κάποιες επαφές με τον Καναδά, συνεχίζονται, αλλά η πρώτη επίσημη, το πρώτο επίσημο βήμα είναι η έκθεση προς την Επιτροπή Εμπορίου. Στο πλαίσιο αυτό θα έχουμε και την Επιτροπή Βιώσιμης ε, Ανάπτυξης, έχουμε συναντήσεις ε, με, τα, με, με, το με την Εσωτερική Συμβουλευτική Ομάδα, κοινέ συναντήσεις όπου θα συζητηθεί το ζήτημα αυτό. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για τα αποτελέσματα αυτά. Τούτο εξαρτάται από το περιεχόμενο. Τώρα συζητούμε το περιεχόμενο της ρήτρα ε, αναθεώρησης. Η επόμενη, το επόμενο ορόσημο, ωστόσο, είναι η έκθεση προς την Επιτροπή Εμπορίου. Δεν έχουμε στη φάση αυτή μία θέση για το τελικό αποτέλεσμα. Συζητούμε ακόμα τις διαδικασίες και την οπτική που θα έχει αυτή η τυχόν ρήτρα αναθεώρησης. Μία επιπρόσθετη ερώτηση από τη συνάδελφο. Να διευκρινίσω για την ενεργοποίηση της ρήτρας διασφάλισης. Ξέρουμε ότι οι χώρες που είναι κάπως λιγότερο αναπτυγμένες δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτή τη ρήτρα γιατί δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για να το πράξουν. Πρώτον. Δεύτερον, συχνά η απόφαση είναι απόφαση των πολιτικών αρχών που δεν λαμβάνουν υπόψη τις αυτό που ζητούν ενδεχομένως τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Για παράδειγμα, εκπρόσωποι των γεωργών που βλέπουν ότι απειλούνται εθνικοί κλάδοι γεωργίας που δεν λαμβάνει όμως η κυβέρνηση υπόψη. Τέτοια αιτήματα που διατυπώνονται στο πλαίσιο των, της επιτροπής που θεσπίζεται στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας επίλυσης διαφορών μπορεί να ληφθεί υπόψη όταν ενεργοποιηθεί η ρήτρα διασφάλισης. Όταν δηλαδή υπάρχουν εθνικές απόψεις που ζητούν κάτι τέτοιο. Συχνά ε, οι ρήτρε διασφάλισης παρουσιάζονται από την Επιτροπή ως ε, πανάκια. Ε, μην ανησυχείτε μας λέτε γιατί υπάρχει ρήτρα διασφάλισης αλλά πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ευκολότερα τέτοιες ρήτρε μετά από θέσεις Τη κοινωνία των πολιτών ή άλλους κλάδους που δεν λαμβάνουν υπόψη οι κυβερνήσει. Αυτό για να διευκρινίσω αυτά που ρώτησε προηγουμένω. Okay. Δεν θέλει να απαντήσει εκπρόσωπος της Επιτροπής. Thank Okay. Ε, ε, να απαντήσω για, το... για κάποιες ερωτήσεις. Μονοπόλιο. Εμείς προτείνουμε το έναν ε, πολύ συγκεκριμένο και διαθρωμένο τρόπο της εσωτερικής συμβουλευτικής ομάδας για να απαντά σε τέτοια αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς είμαστε υπέρ της επέκτασης του μηχανισμού σε όλες τις παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων και των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Σκεφτήκαμε το πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό που κάνουμε. Και εμείς λοιπόν σκεφτήκαμε να σταθούμε σε κάποιες προτεραιότητες. Αν δείτε τις προτεραιότητες στην Κορέα έχετε το πλαίσιο των επικοινωνιών, τα αυτοκίνητα, ε, προδιαγραφές ε, για το προδιαγραφές, άρα πρέπει ο εσωτερικός αυτός ε, συμβουλευτικός ε, φορέας να μπορεί να δει τις απόψεις και προς τα έξω. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά υπάρχουν παρεμπιπτόντως και άλλα βήματα. Εμείς αναφερθήκαμε σε κάποια, σε κάποιους φορείς, αλλά το DAX έχει μια συγκεκριμένη δομή. Τώρα, κυρώσεις δεν είναι δικός μας ρόλος. Ε, από... Δεν θέλουμε να είμαστε δικαστήριο. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Αλλά πρέπει να μπορούμε να, να, να θέσουμε οποιοδήποτε ζήτημα και να παίρνουμε απαντήσεις σε αυτά που θέτουμε. Όταν θέτουμε ερωτήσεις στην Επιτροπή θα θέλουμε να λάβουμε μια απάντηση. Τώρα, εμείς ετοιμάσαμε κάποια κριτήρια για τις διάφορες συμφωνίες. Τις μεγάλες έχουμε δύο μέλη ανά Για τις μικρότερες συμφωνίες ένα μέλος ανά επιτροπή. Έχουμε 69 συμφωνίες. Μιλώ και για τις παλιές που κάποτε θα αναθεωρηθούν. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να το σκεφτούμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τους πόρους να το κάνουμε έχουμε την οικονομική δυνατότητα να το κάνουμε. Ήδη για αυτά που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε θα χρειαστούν περισσότερους πόρου. Αυτό που προτείνουμε είναι η Επιτροπή έχει 3 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια για δραστηριότητε follow follow-up. Σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες καταγγελιών, εμείς θέτουμε το τις απόψεις μας και ελπίζουμε ότι θα μπορούμε να παράσχουμε χρήσιμη σύσταση σχετικά. Προτείνουμε μια πενταετή συμμετοχή με εναλλασσόμενη προεδρία κάθε δυόμιση χρόνια για να μπορέσουν οι διάφορες Τετοιε ομάδε να συναντιούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο με διαφορετικές πρακτικέ εμπειρίε. Αλλιώ είναι η κατάσταση στις ε, χώρε εταίρου. Εμεί σκεφτόμαστε για τον Καναδά που είναι ευκολότερο να έχουμε δύο τέτοιε ομάδε. Η Ιαπωνία έχει μια άλλη προσέγγιση με άλλου εταίρου Η δημιουργία αυτών των εθνικών ε, συμβουλευτικών ομάδων θα είναι δυσκολότερη με κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερική, για παράδειγμα η δουλειά δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που πετύχαμε για τη Χιλή και τις υπόλοιπες χώρες καλό θα ήταν να το κρατήσουμε. Γιατί παίρνει χρόνο να αναπτύξουμε μια τέτοια προσέγγιση. Ελπίζω να μπόρεσα να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Κατά την άποψή μου, θα δείτε η έκθεση περιέχει και άλλες απαντήσεις και άλλες ιδέες. Ευχαριστώ. Πραγματικά το για σκέψη παρέχει η έκθεσή σας. Μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα επιμείνω στα ερωτήματα αυτά για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και πόρους για την δημιουργία αυτών των επιτροπών. Ευχαριστούμε λοιπόν. Κλείνει το σημείο 12. Σημείο 13 ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή των μα... της μακροοικονομικής βοήθειας σε τρίτες χώρες. Την συζήτηση αυτή την είχαμε διεξαγάγει πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις τέτοιας μακροοικονομικής βοήθειας για πολλές χώρες. Μιλάμε για πολλά κονδύλια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε μία γενική επισκόπηση για το τι συμβαίνει με αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Βαλέντσα, τον μόνιμο εισηγητή, θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή, τον κύριο Γκρίσε που είναι ε, αναπληρωτής ε, επικεφαλής της ομάδας ΕΚΦΙΝ και τον κύριο Λένερτ που είναι επικεφαλής του κλάδου. 5-7 λεπτά. Καλημέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πολύ για τη δυνατότητα που μα δίνετε να συζητήσουμε μαζί σα το ζήτημα τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση του πώ έχουν τα πράγματα όσον αφορά τις πέντε, τα πέντε προγράμματα μακροοικονομική χρηματοδότηση ε, που ε, προβλέπονται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ επίση να σα δώσω περισσότερε πληροφορίε όσον αφορά τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, ήδη πληροφορίε από την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε δύο τέτοια προγράμματα για την ε, Ιορδανία και την Τινησία και τρεις στις χώρες τι Αντολικέ: ε, Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία. Δεν προβλέπονται αυτή τη στιγμή τέτοια προγράμματα για τι υποψήφιε ή δυνάμει υποψήφιε χώρε, μολονότι το μέσο αυτό μακροοικονομική και μεταδοτική συνδρομή παραμένει διαθέσιμο αν προκύψουν κρίσει οικονομικέ χώρε αυτέ. Όσον αφορά τώρα την νότια γειτονία, στην Ορδανία έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ με δύο συγκεκριμένε δόσει. Η πρώτη δόση εκταμιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2017, η δεύτερη δόση είναι ακόμα διαθέσιμη και βέβαια θα πρέπει πρώτα να πληρωθούν συγκεκριμένα 11 μέτρα πολιτικής τα οποία έχουμε συμφωνήσει σε μνημόνιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας. Η Ιορδανία έχει σημειώσει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις αυτές κατά τη διάρκεια του 2018. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως το οποίο κρεμεί και το οποίο έχει να κάνει με τις δημόσιες συμβάσεις και ιδίω με τη μεταρρύθμιση του συστήματος προσφυγής για αυτές τις συμβάσεις. Ξέρουμε ότι η Ιορδανία επεξεργάζεται τις σχετικές αυτές μεταρρυθμίσεις και προσβλέπουμε στην έγκριση της σχετικής νομοθεσίας ε, τις επόμενες εβδομάδες. Ξέρετε ότι στο πλαίσιο του προγράμματο αυτού θα πρέπει να σημειώνεται πρόοδο ε, και με το πρόγραμμα του Διεθνού Νομισματικού Τομείου. Αυτό ισχύει και για την ε, Ιορδανία. Προβλέπουμε ότι στην επόμενη διάσκεψη που θα έχουμε για την Ιορδανία, η Ιορδανία θα μα δώσει περισσότερε πληροφορίε. Προβλέπεται στι 28 Φεβρουαρίου μια διάσκεψη στο Λονδίνο για την Ιορδανία και στα μέσα Μαρτίου μια διάσκεψη, η τρίτη στις Βρυξέλλες, όσον αφορά την Ιορδανία και την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, αυτή τη στιγμή εκταμευτούν όλα τα ποσά στα πλαίσια της Μακροοικονομικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής. Μπορούμε να προτείνουμε και ένα νέο πρόγραμμα στην Ορδανία σε σχέση με την κοινή δήλωση που έκανε το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο έχει επισυναυθεί στην αρχική συμφωνία του 2016. Η επόμενη συνεργασία που έχουμε είναι με την Τινησία, ένα πρόγραμμα 500 εκατομμυρίων ευρώ σε τρεις δόσεις. Το πρόγραμμα αυτό, όπως και για την Ορδανία, προβλέπει ότι από τη μία πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί προοδος στα πλαίσια του προγραμματος του διεθνους Νομισματικού Ταμείου και από την άλλη περιμένουμε να εφαρμοστεί μία ακόμα προυποθεση σε σύνολο 8 προυποθεσεων προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκταμείευση της δεύτερη δόση. Ουσιαστικά αναφερόμαστε εδώ πέρα στην ε, ανεξαρτησία διοικητική του ελεκτικού συνεδρίου της χώρας αυτής, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της έγκρισης μιας νέας νομοθεσίας για το ελεκτικό συνέδριο. Το Κοινοβούλιο τη Τινησία επεξεργάζεται την νομοθεσία αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ την όλη αυτή διαδικασία προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκναμείευση τη επόμενη δόση. Τώρα, όσον αφορά τις, την Ανατολική Κοινωνία, ξεκινάμε με την Μολδαβία. Έχουμε ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων ευρώ, όπου εδώ πέρα ε, συνδυάζουμε δάνεια και επιχορηγήσεις οι αρχές της Μολδαβία έχουν αρχίσει να εφαρμόσουν τα μέτρα πολιτικής, τα οποία προβλέπονται στο Μνημόνιο Συμφωνίας. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε εκταμιεύσει ακόμα την πρώτη δόση του προγράμματος αυτού, γιατί από τον Ιούνιο του 2018 οι πολιτικές προϋποθέσεις για το πρόγραμμα αυτό δεν πληρούνταν καθότι είχαμε διάφορες ανησυχητικές εξελίξεις στη χώρα αυτή, όπως η ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κίσιναο η εκταμίευση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής αναστέλλεται μέχρι να πληρωθούν όλες τις απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις. Όσον αφορά τώρα τη Γεωργία, εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έγκριναν οι συνομοθέτες τον Απρίλιο του 2018. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει έως 45 εκατομμύρια ευρώ, πάλι ένα συνδυασμό επιχορηγήσεων και δανείων υπεγράφει ένα μνημόνιο συμφωνία με μια κάποια καθυστέρηση, καθότι έγινε ανασχηματισμό τον Ιούνιο-Ιούλιο στην χώρα αυτή, αλλά τελικά αποφασίστηκε στι 31 Αυγούστου του 2018 να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο συμφωνία. Μετά την κοινοβουλευτική έγκριση, προχωρήσαμε στην εκταμείευση των 20 εκατομμυρίων ευρώ, τη πρώτη δόση δηλαδή, το Δεκέμβριο του 2018 και σχετικέ πληροφορίε διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις 4 Δεκεμβρίου. Η Γεωργία επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή την εφαρμογή των συγκεκριμένων συνδικών πολιτικής προκειμένου να υπάρχει η δεύτερη δόση των 25 εκατομμύριων ευρώ και προβλέπουμε ότι θα γίνει μια αποστολή παρακολούθηση των εξελίξεων των, την Άνοιξη. Η Γεωργία έχει σημειώσει πολύ θετική πρόοδο στα πλαίσια του προγράμματο με το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και όλε οι εξολογήσει και των τριών προγραμμάτων ολοκληρώθηκαν εγκαίρω. Τέλος, έχουμε εκταμιεύσει την πρώτη δόση στα πλαίσια της νέ, του νέου προγράμματος μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής με την Ουκρανία, η πιο σημαντική απόφαση τη χρηματοδότησης που έχει ληφθεί από τους νομοθέτες ήδη από τον Ιούλιο του 2018. Προβλέπεται ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε δύο δόσεις. Έντονε διμερεί διαπραγματεύσει έλαβαν χώρα το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το μνημόνιο συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ουκρανία να μπορεί τελικά να υπογραφεί στι 14 ε, Σεπτεμβρίου του 2018 οι προϋποθέσεις για την υποβολή, την εκμεταμίευση της πρώτης δόσης είχαν να κάνουν με την πολιτική διαδικασία στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας. Η Ουκρανία κατάφερε να καλύψει και τις έξι δεσμεύσεις πολιτικής, προκειμένου να έχουμε την πρώτη δόση στα μέσα Νοεμβρίου περίοδο κατά την οποία τελικά επικυρώθηκε και η σχετική νομοθεσία από το Κοινοβούλιο. Εδώ προβλέπονται συγκεκριμένε μεταρρυθμίσει για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Για πρώτη φορά προβλέπεται ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την δήλωση του πόστου θα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων στη χώρα. Αυτό ήταν η σημαντική απέτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρετε στο παρελθόν είχε οδηγήσει στην ε, ακύρωση της τελευταίας δόσης του προηγούμενου προγράμματος MFA. Η Ουκρανία επίσης άλλαξε τη διαδικασία εταιρικών μητρών προκειμένου να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους συγκεκριμένων επιχειρήσεων και αυτό αποτελούσε προϋπόθεση που δεν είχε καλυφθεί στο παρελθόν. Επίσης, εξίσου σημαντικό, η χώρα ενέκρινε νέο σύστημα διορισμού δικαστών στον Νότο Δικαστήριο Καταπολέμησης της Διαφθοράς. Κατά αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να εκταμιεύσει την πρώτη δόση των 500 εκατομμύριων ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018 και οι σχετικές πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 30 Νοεμβρίου, όπου προβλέπεται μία λεπτομερής ανάλυση των έξι βασικών προποθέσεων. Εν γέννη όσον αφορά λοιπόν την Ουκρανία μετά από μια αρχική επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων του 2016-2017 βλέπουμε τώρα η χώρα σημειώνει εκ νέου πρόοδο, έχει επιταχύνει τι μεταρρυθμίσει τη, ανταποκρίνεται στις δεσμεύσει τη και κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει και πιο έντονη διεθνή υποστήριξη τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο όμω και από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο που το Δεκέμβριο του 2018 ανέκρινε ένα νέο πρόγραμμα για τη χώρα, αλλά υποστήριξη έχουμε και από την Παγκόσμια Τράπεζα, υποστήριξη που υπεγράφει τον Δεκέμβριο. Η ε, Ουκρανία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να προτιμάσει τις, προετοιμάσει, τις μεταρρυθμίσεις για τη δεύτερη δόση. Τον επόμενο μήνα θα πάμε στην Ουκρανία και αν όλα εξελιχθούν ε, θετικά και με το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα προχωρήσουμε στην εκταμείευση της δεύτερης δόσης στην Άνοιξη. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας και εγώ αλλά και ο συναδελφός μου παραμένουμε στη θέση σας για τυχόν ερωτήσεις. Βαλές έχει το λόγο. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή η χρηματοοικονομική αρρωγή ε, προς την Ουκρανία ε, από το 2014 έχει φτάσει στα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ οπότε πρόκειται για τη μεγαλύτερη αρρωγή που έχουμε παράσχει σε ε, χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τώρα, η πρόταση που ήρθε στα τέλη του Νοεμβρίου ήρθε σε μια πολύ κέρια χρονική συγκυρία γιατί οι άνθρωποι της Ουκρανίας αντιμετώπιζαν μια κλιμάκωση της σύγκρουσης και μια αύξηση της απειλής βάρος τους στη θάλασσα του Αζόφ. Οπότε πραγματικά πρόκειται για πολύ σημαντικό σημαντική χρονική συγκυρία. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Ουκρανία ανταποκρίνεται στι δεσμεύσει που έχει αναλάβει σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει τη ε, παρά το ανασφαλέ περιβάλλον. Θα πρέπει δηλαδή θα πρέπει να θυμηθούμε τι επερχόμενε προεδρικέ εκλογέ, τι επερχόμενε κοινοβουλευτικέ εκλογέ, οπότε γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε κυβερνητικό επίπεδο όταν επίκυνται εκλογές. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η Ουκρανία καταφέρει να ανταποκριθεί σε μία σειρά από τις που έχει αναλάβει σε επίπεδο πολιτικής ε, και εκεί περιλαμβάνονταν για παράδειγμα επίτευξη των μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αύξηση της διαφάνειας των εμπορικών των μικρών επιχειρήσεων και προβλεψιμότητα του φορολογικού πλαισίου, καθώς και ενίσχυση της διακυβέρνησης ε, και της δυνατότητας διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων. Και εμείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης ε, πράγματα πρέπει να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην συνέχιση αυτών των προσπαθειών, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά και τον, τα μέτρα σε επίπεδο δικαστικό σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ωστόσο εδώ δράτω με τις ευκαιρίες για να θέσω κάποια ερωτήματα σε ό,τι αφορά κάποια εμπόδια στο εμπόριο τα οποία παραμένουν. Ε, καταρχήν, σε ό,τι αφορά την άρση της απαγόρευσης εμπορίου ε, ξυλίας ε, που ισχύει από το 2015 και η οποία έρχεται σε αντίθεση με το γράμμα και το πνεύμα της ε, συμφωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά την διαφάνεια των εγγράφων σε σχέση με τις εξαγωγές παλιοσιδέρων, θα ήθελα να μας ενημερώσετε περισσότερο. Τέλος, θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές επουλερικών υπό τον κώδικο της συνδεδεσμένης ε, ονοματολογίας 0207-1370. Γιατί εκεί χρησιμοποιείται ουσιαστικά ο κωδικός ε, για άλλα ε, μέρη, αν θέλετε, πουλερικού, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για στήθος Κοτόπουλου. νομίζω πως εδώ δεν ακολουθούμε το όσο προβλέπει η συμφωνία και δημιουργεί ένα παραθυράκι, αν θέλετε, ένα ε, ένα είδο καταστρατήγηση σχετική ε, συμφωνία. Ε, δημιουργεί δηλαδή μειονεκτική θέση για του δικού μα παραγωγού και ουσιαστικά πρόκειται για ένα σημείο που έχει υπάρξει δημιουργική εντό εισαγωγικών η πλευρά τη Ουκρανίας. Θα ήθελα κάποιες απαντήσεις σε σχέση με αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σούστερ έχει το λόγο, λέει ο πρόεδρος. Ναι, θα συμφωνήσω πλήρω με τα όσα είπε μόλι τώρα ο κ. Βαλέσσα. Δηλαδή, την τελευταία φορά είχαμε συζητήσει επί μακρόν κατά πόσο θέλουμε πράγματι να συνεχίσουμε την ε, χορήγηση της ε, χρηματονομικής αρρωγή ε, προς την Ουκρανία και τότε είχαμε πει ότι πριν ακόμα καταβάλουμε προκαταβολές θα πρέπει να ε, ενημερωνόμαστε ως προς το πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιωθεί ο όλος ο ε, πολύ περισσότερο. Δηλαδή δεν θα πρέπει απλώ κάποια στιγμή να βλέπουμε ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρει εκταμίευση τέτοιου είδου ε, αρρωγή. Από εκεί και μετά. Θα ήθελα να μα πει η Επιτροπή τι ακριβώ ε, θεωρεί πω αποτελεί βελτίωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή και την καταπολέμηση τη διαφθοράς. Γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ουσιαστικά εγκαταλείπουν τη χώρα, από, οι πλούσιοι δηλαδή ουσιαστικά τα κάνουν να φύγουν από τη χώρα και είναι πολύ ψηλότερα αυτά τα κοντήλα από αυτά τα οποία εισέρχονται στην Ουκρανία από τη δική μας πλευρά. Δηλαδή τελικά ο απολογισμός ε, δεν ξέρω αν είναι θετικός. Οπότε ποιο είναι το κριτήριο τελικά με βάση το οποίο μας λέτε ότι λαμβάνει η χώρα ε, κατά πολέμηση της διαφθοράς. Γιατί εγώ δεν γνωρίζω καμία υπόθεση σημαντική όπου ε, υπήρξε μια υπόθεση που βρέθηκε ενώπιον δικαστηρίου και πολύ λιγότερο βέβαια να έχει καταδικαστεί κάποιος. Η ε, ολιγαρχία δηλαδή αυτή η λίγη αν θέλετε ιδιαίτερα εύποροι πολίτες συνεχίζουν ε, την δραστηριότητά τους ως ε, έχουν και κανένας δεν φοβάται από ό,τι φαίνεται να απολέσει την περιουσία του. Οπότε για μένα είναι θεμελιώδες αυτό το ερώτημα. Τι ακριβώς σημαίνει καταπολέμηση της διαφοράς για την Ευρωπιτροπή. Γιατί δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι ουσιαστικά ε, για πολιτικούς λόγους η Επιτροπή λέει ότι ό,τι και αν γίνει θα πρέπει να ε, συνεχίζουμε να επενδύουμε, αν θέλετε, λεφτά σε αυτή την ε, χώρα. Ε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ουσιαστικά συμβαίνει αυτό, δηλαδή να υπάρχει συνεχώς υποστήριξη από τη δική μας πλευρά, αλλά η Ουκρανία δεν ανταποκρίνεται σε κάτι, δεν αλλάζει κάτι εκεί και η Επιτροπή παρόλα αυτά συνεχίζει να υποστηρίζει ε, χρηματοοικονομικά αυτή τη χώρα. Οπότε θα ήθελα η Επιτροπή να μα πει πώ θα συνεχίσει να μα ενημερώνει ε, το Κοινοβούλιο, όχι μέσω απλώ δελτίων ε, τύπου, ή προκαταβολικά έκτο των προτέρων πώς θα μα ενημερώνει από εδώ και στο εξή. Πώ λοιπόν σκοπεύει να το κάνει αυτό, και το δεύτερο ερώτημα, όπω το είπα, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό είναι τι ακριβώ θεωρεί πω λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία για να θεωρήσει πω υπάρχει καταπολέμηση τη διαφθορά. Πώ αντιλαμβάνεται την καταπολέμηση τη διαφθορά. Παρακαλώ. Ένα ακόμα μιλητή. Ναι, ε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη συζήτηση που γίνεται για την Ουκρανία, όπως είχε ε, γίνει πέρσι, ότι δηλαδή είχε τεθεί ε, πίεση στο, είχε ασκηθεί πίεση στο Κοινοβούλιο, ως προς το να δεχτεί τη σχετική συμφωνία και να μην φέρει αντίβηση σε ό,τι αφορά τις Βασικέ διατάξει τη συμφωνία. Οπότε για μας ε, είναι πολύ σημαντικό αυτέ οι διατάξει να τηρούνται και να πληρούνται και όπως αυτές συναντεύουν τη χρηματοοικονομική αρρωγή. Να πω λοιπόν σχετικά ότι είναι θετικό το γεγονό ότι βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Ωστόσο, αυτή η έναρξη των μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί επίτευξη του σχετικού στόχου. Δηλαδή, ο στόχο σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το δικαστήριο και την καταβολή τη διαφθορά, ε, ο στόχο ο πραγματικό είναι να αναλάβει κανονικά δραστηριότητε, να, να, να, να ξεκινήσει τι εργασίε του αυτό το δικαστήριο. Μετά, σε ό,τι αφορά ε, τι μεταρρυθμίσει, αυτέ θα πρέπει να είναι βιώσιμε και α, ε, κοινωνικά. Ε, θεμητές. Είναι θετικό το ότι έχουν ξεκινήσει κάποιε μεταρρυθμίσει, αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερο ω προ το πώ ακριβώ. Ε, θα επιτευχθεί με αυτού του στόχου μια ανάπτυξη χωρί ε, αποκλεισμού και ειδικότερα πώ διασφαλίζεται ο ρόλο τη κοινωνία των πολιτών. Επίση, στο ενημερωτικό σημείωμα υπάρχει μια παράγραφο η οποία αναφέρεται στην πρώτη συμφωνία χρηματοοικονομική αρρωγή. Και εκεί αναφέρεται λοιπόν ότι παραμένουν μια σειρά από ανησυχίε σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί έναν από του βασικού πυλώνε μια τέτοια συμφωνία χρηματοοικονομική ε, αρρωγή. Οπότε, με ποιον τρόπο ε, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας η Επιτροπή ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανησυχίες, ε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι πραγματικά είμαι πολύ θετικός απέναντι, θετικά διακείμενος απέναντι στην Ουκρανία και στην υποστήριξη του λαού της, γιατί πρόκειται για μια σημαντική γειτονική χώρα. Ωστόσο, η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει ε, ένα πραγματικά υψηλά ποσά και γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να λάβει υπόψη της όλα τα επιμέρους ζητήματα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο λόγος τώρα στην Επιτροπή για να απαντήσει όλα αυτά τα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ. Ξεκινώ. Προβλήματα στο εμπόριο. Πρώτα πρώτα να σας διευκρινίσω ότι εμείς είμαστε από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ κάποιο συνάδελφο από την εμπορική διάσταση. Μπορώ να σα πω λοιπόν αυτά που ξέρω που σχετίζονται με την σύνδεση που κάνουμε μεταξύ εμπορικών διαστάσεων και μακροοικονομικής βοήθειας. Ε, φαντάζομαι ότι αυτό θα εμφανίζεται σαφώς στο τρίτο πρόγραμμα μακροοικονομικής βοήθειας. Όπως ε, σας είπε, όπως ξέρετε, στην πρότασή της για, το τέταρτο, για την τέταρτη σχετική απόφαση, η Επιτροπή δεν προτίθεται να συμπεριλάβει την απαγόρευση εξαγωγής ε, ξυλίας στο τέταρτο αυτό πρόγραμμα μακροοικονομική βοήθεια, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημα συγκεκριμένα εξειδικευμένα εμπορικά εργαλεία. Προ το παρόν μπορώ λοιπόν να επιβεβαιώσω μόνο ότι ο οργανισμός ε, ε, επίλυση διαφορών με βάση την συμφωνία με την Ουγγαρία έχει ε, ενεργοποιηθεί και ορίστηκαν τα άτομα. Ειδικά για την απαγόρευση εξαγωγή ξυλία οι πρώτε διαβουλεύσει για το σημείο, επίσημε διαβουλεύσει για το για το θέμα αυτό με βάση το DCFTA θα ξεκινήσουν αρχές Φεβρουαρίου. Ξεκίνησαν αρχέ Φεβρουαρίου, συγγνώμη. Ανάλογα με την έκβαση των διαβουλεύσεων θα αποφασιστεί κατά πόσον μία από τα, ένα από τα δύο μέρη, η Ένωση στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα παραμπέψει επίσημα το ζήτημα αυτό στο μηχανισμό επίλυσης διαφορών για το σκραπ ε, σιδερικών και τα ε, στήθη πουλερικών. Δυστυχώς δεν έχω πληροφορίες, θα παραπέμψω το θέμα στον συνάδελφο που ξέρει το ζήτημα αυτό. το ζήτημα για τις απαιτήσει ενημέρωσης. Η απόφαση για τη μακροοικονομική βοήθεια εγκρίθηκε από τους συνομοθέτες αρχές Ιουλίου. το καλοκαίρι διαπραγματευτήκαμε το μνημόνιο συνεννόησης. Τέλη Αυγούστου, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά γύρω στις 24 Αυγούστου υποβλήθηκε το σχέδιο μνημονίου συνεννόησης το Μητρό Επιτροπολογίας. Τα κράτη-μέλη κλήθηκαν σε μια συνεδρία της Επιτροπής που έγινε στι 6 Σεπτεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε πήρε πρόσβαση στο κείμενο του σχεδίου μέσω του Μητρώου ε, Επιτροπολογίας που ρυθμίζεται από τον κανονισμό ε, επιτροπολογίας που έχει σχεδόν ιονή ε, συνταγματικό χαρακτήρα και μας θέτει μια σειρά υποχρεώσεων. Οπότε από τα τέλη Αυγούστου έχετε το σχέδιο του μνημονίου όλοι. Κατόπιν υπογράφηκε 14 Σεπτεμβρίου και υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή με τα κρατη 6 Σεπτεμβρίου και υπογράφηκε στις 14. Έκτοτε είναι δημόσιο έγγραφο. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, δυνατότητα όλοι να δουν το κείμενο αυτό στην ιστοσελίδα μας. Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση. Όντως βγήκε ένα ανακοινωθέν τύπο από εμά, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο κείμενο που δώσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας στείλαμε και ένα ενημερωτικό σημείωμα 20, 20 σελίδες περίπου με μια λεπτομεριακή ανάλυση όλων και των έξι δηλαδή προϋποθέσεων που συνδέονται με την πρώτη εκταμείευση καθώς και ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΔΝΤΑΦ. Υπάρχει λοιπόν διαφάνεια και είναι σαφές νομίζω σε όλους γιατί θεωρούμε ότι τηρήθηκαν οι προποθέσει για αυτή την εκταμείευση με βάση και την κοινή δήλωση δημοσιοποιήσαμε το κείμενο αυτό στην ιστοσελίδα μας γιατί και σε αυτό δεσμευτήκαμε. Ε, ε, σε ό,τι αφορά την πρόοδο στην καταπολέμηση διαφθοράς και της ε, φόρο διαφυγής αναφέρατε ότι δεν είδατε να καταδικάζεται από τα δικαστήρια κάποιος Ουκρανός πολιτικός επιχειρηματίας. Βεβαίω, όταν κοιτούμε τη μακροοικονομική βοήθεια πρέπει να δούμε τι συγκεκριμένες δράσεις μπορεί να συμπεριληφθούν ε, στους όρου τη εκταμίευσης. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα πρόγραμμα μακροοικονομικής ε, βοήθεια ότι η Ουκρανία δεσμεύεται να καταδικάσει ένα χι αριθμό απαταιώνων. Δεν μπαίνουν κάτι τέτοια. Πρέπει να αναφέρουμε τις θεσμικές ή άλλες μεταρρυθμίσεις που υλοποιούν τις απαιτήσει ούτω ώστε κάτι τέτοιο να γίνει στο μέλλον. Όπως σας είπα το μνημόνιο συνεννοήσεις είναι δημόσιο και μπορείτε να δείτε τι θεωρούμε ως πρόοδο και ότι αυτό που θεωρούσαμε ως πρόοδο ήταν επαρκές για να εκταμιευθεί το συγκεκριμένο κονδύλι. Υπήρξαν μια σειρά δηλώσεων δημοσίων αξιωματούχων. Το κείμενο είναι σημαντικό. Ε, μπορείτε να συγκρίνετε τι δηλώνει ο κόσμος, είτε τα οι επιχειρηματίες και οι πολιτικοί σε σχέση με το τι λαμβάνουν. Υπάρχουν δηλαδή μια σειρά μηχανισμών ε, διαπίστωση του κατά πόσον το πόθεν έσχεση των πολιτικών είναι ε, πραγματικό ή όχι. Αν ξέρει ότι πρέπει να δηλώσει την περιουσία σου όταν εκλέγεσαι ω βουλευτή ή αποκτά μια θέση στην κυβέρνηση και έχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ, μπορεί να μην, το, να μην κατέβεις υποψήφιος και αυτό είναι κομμάτι της καταπολέμησης διαφθοράς. Τώρα το δικαστήριο που, αυτό το δικαστικό όργανο που θα αντιμετωπίζει την διαφθορά. Ε, έκανα μια σχετική αναφορά στις αρχικές παρατηρήσεις μου. Υπάρχουν υποχρεώσεις που δεν αποτελούν πανάκια για την επίλυση όλων των προβλημάτων της Ουκρανίας βεβαίως, αλλά υπάρχει σίγουρα πρόοδος προς κάποια, κάποιες κατευθύνσεις. Αν δείτε την κατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μη σας πω της Ένωσης, θα δείτε ότι η μάχη κατά της διαφθοράς πάντα είναι δύσκολη. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει υποχώρηση. Και βέβαια, τους όρους αυτούς, τους παρακολουθούμε, τις προϋποθέσεις αυτές παρακολουθούμε προσεκτικά όταν ετοιμάζουμε μία απόφαση εκταμίευσης και δείξαμε σαφώς ότι τέλη 17, 18 δεν εκταμιεύουμε χωρίς προϋποθέσεις. Η τελευταία εκταμίευση του τρίτου προγράμματος δεν εκταμιεύτηκε διότι δεν είχαν εφαρμοστεί κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις. Αυτό το μήνυμα το κατάλαβαν και στην Ουκρανία. So um, then maybe briefly turning to uh, the question regarding Τώρα, Ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στις κοινωνικές διαστάσεις και την ε, ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Θα δείτε ότι υπάρχουν ε, στο μνημόνιο συγκεκριμένοι κανόνες ε, κοινωνικής ανάπτυξης για την εκταμίευση της δεύτερης δόσης, χρηματοδότηση της περίθαλψης, συγκεκριμένη στοχοθέτηση των κοινωνικών επιδομάτων, ενίσχυση και βοήθεια στους εσωτερικά διοχθέντες. Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών και ολόκληρη της συμφωνίας δηλαδή ε, που εμφανίζεται στο ενημερωτικό σημείο του Μνημόνιου Συνεννόησης δείχνει την κατάσταση. Ξέχασα να σας πω, έπρεπε να σας το είχα πει ότι δεν δώσαμε μόνο το σχέδιο μνημονίου, αλλά δώσαμε και ένα background note για το γιατί επιλέξαμε συγκεκριμένες πολιτικές, ποιος ήταν ο αντίκτυπος και θα υπάρχει και ένα, και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο σε αυτό το ιστορικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο σε όλους. αναφερθήκατε και στο δικό μας ε, σημείωμα για την πρώτη εκταμίευση. Μιλήσατε για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δική μας ε, εκτίμηση είναι ότι οι πολιτικές προϋποθέσεις ε, στην Ουκρανία πληρούνται. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου που αφορούν κυρίως, τον, αφορούν κυρίως τον, τα εδάφη που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση ό,τι αφορά τον χώρο που ελέγχει η κυβέρνηση, τα, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι παρκής Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Βαλένσα και Σούστερ. Ε, δεν έχει νόημα να θέσω ερώτημα. Απλώς διαπιστώνω ότι δεν είναι επαρκές ε, να γίνεται μια ενημέρωση όπως αυτή έγινε μόλις τώρα. Δηλαδή ε, οι ευρωβουλευτές μπορούν να ρίξουν μια ματιά στην ιστοσελίδα μας. Ε, δεν πρόκειται για ενημέρωση σωστή, ειδικότερα όταν πρόκειται για πολιτικά αμφιλεγόμενα ζητήματα. Και από εκεί και μετά δεν νομίζω πως επαρκεί να διαπιστώνουμε κατά πόσο υπάρχουν κάποιε επίσημε θεσμικέ δομέ. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα τη φοροδιαφυγή και τη καταπολέμηση τη διαφθορά, η ίδια Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει ε, ή να, να βεβαιώνεται ότι πραγματικά καταπολεμάται στην πράξη φοροδιαφυγή. Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και καιρό. Οπότε, επειδή ακριβώ δεν έχει υπάρξει δίωξη μέχρι τώρα, ε, ε, θα πρέπει να το εξετάζει πολύ προσεκτικά η Επιτροπή το να δημιουργούνται δηλαδή κάποιες δομές οι οποίες ε, απλώς και μόνο ενδεχομένως ε, ε, ονομαστικά υπάρχουν για την καταπλήρωση τη διαφορά, χωρίς όμως να έχουν αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να επαρκεί για την Επιτροπή και δεν θα πρέπει να επαρκεί για μας. Ευχαριστώ. Ο κύριο Βαλέζα, θα ήθελα να ζητήσω γραπτή απάντηση στι ερωτήσει μου, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε, ιδίως για τα όσα είπατε για το εμπορικό τμήμα. Θα έχετε μια γραπτή απάντηση και έχουμε και την δήλωση του κύριου Χιουστέρ, η οποία εξακολουθεί να ισχύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί και έχει εδώ πέρα κάποιες υποχρεώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται έτσι και το σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης και μπορούμε έτσι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση των συντονιστών σε ένα λεπτό. Κάνουμε διάλειμμα ενός λεπτού και όσοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν, ας αποχωρήσουν.